Proszę Państwa, otwieramy posiedzenie naszej komisji. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το σημείο 20. Μία έκθεση για την συνεδρία των συντονιστών. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής. Οι συντονιστές επιβεβαίωσαν ότι δεν θα υπάρξουν ε, επιπλέον επισκέψεις της Επιτροπής μας κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Δηλαδή από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ισχύει αυτό. Επίσης, Επιβεβαιώνουμε την απόφαση που πήρε χθε η Επιτροπή, επιβεβαιώσαμε ως συντονιστές. Ζητάμε δηλαδή την έγκριση του Κοινοβουλίου για την έκθεση Μαρτίνας Μαρτίνας για την ειδική έκθεση του διαμεσολαβητή για τους διερμηνείς ACI. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρότι λοιπόν είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα εξετάσουμε επιπλέον ε, εκθέσεις, ζητάμε την άδεια του Κοινοβουλίου να εξετάσουμε αυτή την έκθεση και μόνο του διαμεσολαβητή. Επίσης, είπαμε ότι η έκθεση Μαγκίνες για τις ετήσιες δραστηριότητές μας θα ψηφιστεί στην Επιτροπή στις 31 Μαρτίου. Στην συνεχεία ανταλλάξαμε απόψεις εν ώψη της έκθεσης Χάμενστάιν Μίντσε. Εν συνεχεία, κοιτάξαμε τον κώδικα καλών πρακτικών που ετοίμασε η ομάδα του ΕΛΚ της Επιτροπής μας με συμφωνία με τους σοσιαλιστές, σε συμφωνία με τους σοσιαλιστές. Συμφωνήσαμε ότι το έγγραφο αυτό θα μεταφραστεί στις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής και στις συνεδρίες που θα κάνουμε στις 31 Μαρτίου θα συζητήσουμε το έγγραφο και θα το υιοθετήσουμε αν γίνεται. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν ή όχι επίμαχα σημεία. Ο Σερ Ρόμπερτ όμως ζήτησε να μπει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ε, της 31ης Μαρτίου και θα ασχοληθούμε με αυτό το κείμενο 20 λεπτά. Εάν μπορούμε σε 20 λεπτά να το διεκπαιρεώσουμε και να το υιοθετήσουμε, έχει καλό. Αλλιώς θα δούμε αργότερα τι μπορούμε να κάνουμε το λόγο κείμενο. Οι συντονιστές Θα ήθελα να υιοθετηθεί αυτός ο κώδικας διοντολογίας, αυτός ο κώδικας καλών πρακτικών, πριν λήξει η θητεία του Κοινοβουλίου. Αυτά έχω να σας πω λοιπόν από την ε, συνεδρίαση των συντονιστών και τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Σύνοτ για τον ενεργό διάλογο με τους πολίτες με θέμα την Ευρώπη. Εν συνεχεία θα ψηφίσουμε την έκθεση ΑΟΚΕΝ Ένα διαδικαστικό πριν περάσουμε στην έκθεση Auken που θα είναι μια δύσκολη έκθεση στην ψηφοφορία όπως ξέρουν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι ζήτησα εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ με την υποστήριξη άλλων συντονιστών από άλλες ομάδες να υιοθετήσουμε τη βάση του άρθρου 178 σε ό,τι αφορά τους ε, συναδέλφους θα ψηφίσουν και τους αναπληρωτές. Υπάρχουν 14 μέλη του ΕΛΚ, 12 ε, σοσιαλιστές, 3 φιλελεύθερους, 3 ΟΕΝ, 3 πράσινοι και ένας ανεξάρτητος. Και ένας μη εγγεγραμμένος. Αυτό είναι το σύνολο. Σας κοινοποίησαμε, Πρόεδρε, και και οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι για αυτές τις αλλαγές τους αναπληρωτές. Και πριν γίνει η ψηφοφορία θα ήθελα είτε εσείς ή οποιοδήποτε άλλος να μας επιβεβαιώσετε τον ακριβή αριθμό και, ονο... και όνομα του αναπληρωτή που θα ψηφίσει. Για αυτό το θέμα, την έκθεση Άουκεν πάντα, έτσι. Δεν θα είμαι ο συντονιστής του ΕΛΚ, αλλά η κυρία Ντεκόν θα είναι η συντονίστρια γιατί εγώ θα έχω μια κατάλληλη διαφορετική θέση. Κύριος ε, Κάσμαν. Ο κύριος Πόπα θα είναι σήμερα το πρωί εδώ. Δεν ξέρω αν αλλάζετε τη δήλωσή σας για το, τους συντονιστές. Πάντως πριν από την ψηφοφορία θα ελέγξουμε ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι αναπληρωτές έχουν ενημερωθεί. Σε Ρόμπερτ. Ο κύριος Πόπα από δεν θα είναι εδώ. Αλλά αν είναι εδώ πρέπει να έρθει γρήγορα. αν είναι έρθει θα είναι. Θα πρέπει να έρθει γρήγορα. Ε, αν έρθει, ε, έχει καλώς. Αν, αλλιώς η κυρία Ντεκάν θα ψηφίσει τη θέση του. Ο κύριος Χάμερστάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθούμε στο κεφάλαιο, έρθρο, 1 ε, του, το άρθρο 108 του κανονισμού του σώματος όπου λέει σε περίπτωση απουσίας ενός τακτικού μέλους το τακτικό μέλος της Επιτροπής είναι δυνατόν να αντικατασταθεί στις συνεδριάσεις από άλλον βουλευτή της ίδιας πολιτικής ομάδας, ο οποίος θα έχει δικαίωμα ψήφου το τακτικό μέλος θα πρέπει να γνωστοποιήσει το όνομα του αναπληρωτού στον πρόεδρο. Μία πολιτική ομάδα δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο αριθμό αναπληρωματικών μελών από ό,τι τακτικά μέλη. Θα ήθελα να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός όσον αφορά τη διαδικασία ψηφοφορίας. Παρακαλώ να εγγραφεί στα πρακτικά. Thank uh, um, Ευχαριστώ. Έχω ένα αντίγραφο του κανονισμού μπροστά μου και η γραμματεία θα εφαρμόσει αυτό το κανονισμό πριν την ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι, θα είναι μια δύσκολη ψηφοφορία. Θα, θα σας βοηθήσω αν με βοηθήσετε. Σας παρακαλώ να μην γίνετε ψήφιρο στο... και συζητήσει στο βάθος. Αν δεν υπάρχουν ψήφιροι φασαρίες, συζητήσεις, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία και πρέπει να είμαστε ακριβείς. Σας παρακαλώ, δείξτε λίγη κατανόηση και βοηθήστε τον εαυτό σας και όλους μας για την ψηφοφορία. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα Με ακούτε στο βάθος. Εγώ σας ακούω. Αυτό είναι το θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Σίνατ να κάνει μια δήλωση πριν ψηφίσουμε. Και αν δεν έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, στείλτε κάποιον σας τις φέρει, παρακαλώ, κυρία Σίνατ. Ένα σύντομο σχόλιο για τον κατάλογο ψηφοφορίας. Η έκθεση έχει ένα απλό μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι όταν επικοινωνεί κανείς με τους πολίτες, οι ε, πράξεις είναι πιο εύγλωτες από τα λόγια. Και η πράξη που θα ήθελα να υπάρξει, να προωθηθεί στην έκθεσή μου, είναι να δώσουμε περισσότερους πόρους σε αυτή την Επιτροπή, ούτως ώστε να μπορούμε να ενεργούμε ε, εκ μέρου των πολιτών και για τους πολίτες. Είναι απλό μήνυμα. Ε, και ορισμένε τροπολογίες το απεικονίζουν αυτό το μήνυμα. Ε, υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που δεν το απεικονίζουν και δεν υπάρχουν εδώ. Ε, εσείς τα αποφασίσετε. Ε, αν αυτό το μήνυμα φύγει, δεν έχει νόημα καθόλου η έκθεση. Αυτή είναι η σύστασή μου. Σας παρακαλώ να παραμείνει αυτό το μήνυμα θα μπορούσαμε να πούμε στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που χρηματοδοτούν ε, και επανδρώνουν αυτή την Επιτροπή. Κύριος Κάσμαν, ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να μιλάω πιο δυνατά από εκείνους που ψιθυρίζουν και μιλάνε στην αίθουσα. Θα ήθελα να ενημερώσει κάποιο του ανθρώπου που μπαίνουν ότι θα πρέπει να μπαίνουν σιωπηλά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί το σύστημα, ότι τα νούμερα είναι σωστά. Ψηφίστε ελεύθερα, ψηφίστε όπως θέλετε, αλλά ξεκινάει η ψηφοφορία. Ησυχία παρακαλώ. Uh, David. I think would be, it would be good to know who are, who are the voting Νομίζω ότι καλό θα ήταν να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα ποιοι έχουν δικαίωμα ε, συμμετοχή στην ψηφοφορία. Κοιτάξτε, ελέγχεται αυτό. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και ταυτίζουμε τα ονόματα με τους παριστάμενους, με τα πρόσωπα. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο πράγματι λειτουργεί αυτό το ε, ηλεκτρονικό σύστημα ψηφορίας. Άρχεται η ψηφορία, παρακαλώ να ψηφίσετε. Έκλεισε. Ψήφισαν 35 από τους 36. Αν έχετε την καλοσύνη να δούμε στην οθόνη το αποτέλεσμα. Okay, if we can vote once. Λοιπόν, ε, ξαναψηφίζουμε. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Έκλεισε. Το πρόβλημα είναι ότι ψήφισαν 36, αλλά εμείς στον κατάλογό μας έχουμε μόνο 33 ονόματα. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε ο κύριος Κασπάρη είναι παρόν. Ο κύριος Κασπάρη, ο κύριος Κόρμπιτ. If you bear with us, it's extremely important that we get this settled before any votes are taken. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να δείξετε κατανόηση, πρέπει να το ρυθμίσουμε το θέμα πριν αρχίσουμε την καταμέτρηση των ψήφων.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 δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε παρέμβαση θα βοηθούσε. Μισό λεπτό περιμένετε. Okay, this is, um, ladies and gentlemen, this is what I'm Κοιτάξτε, θα πρέπει δυστυχώς ε, να συνεχίσουμε με ονομαστική ψηφορία. Δηλαδή, ε, θα ζητήσω ποιοι είναι παρόντες, ε, εάν είναι εδώ, παρακαλώ να το δηλώνουν και αν δεν είναι παρόντες όσοι θα ακούν το όνομά τους, να μας το επισημαίνουν οι αναπληρωτές τους για να τσεκάρουμε τον κατάλογό μας. Λοιπόν, είναι καλύτερα να ακούτε ονόματα στο πρωτότυπο. Yes. Thank you. Um, David Martin. Thank you. Uh, Miguel Martinez. Thank you. Um, replaces is replacing uh, Maria Matsuka. Yáñez? No, yet? yes. Pardon. Um, Mr. Mavromatis? Thank you. Uh, Mr. Meyer? Thank you. Uh, uh, Mr. Mitchell?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 Mr. Battilaccio? Yes. Mr. Thomas. Mrs. Tomaszewska. Mrs. Tomaszewska. Thank you. Mr. Uh, Mr. Busitil. Thank you. Michael Cashman, yes. And Jules Martin, representing Mr. Costa. Thank you. Riera. Riera, representing De Rosa.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 So and anyone who has not been called, ladies and gentlemen, anyone who has not been called cannot. Υπάρχει κάποιο που δεν άκουσε το όνομά του, γιατί αν δεν άκουσε το όνομά του είναι προφανέ ότι δεν μπορεί να ε, ψηφίσει. Αν ε, δεν έρθει ο κύριο, εκτό αν ο κύριο Κάσπαρη ε, έρθει προφανώ την κατάλληλη στιγμή. ο, ε, Τη σωστή στιγμή μάλλον. Λοιπόν, δεν θα ψηφίσουμε, μάλλον ψηφίζουμε για την έκθεση Σύνοτ για το εδάφιο Α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοιτάξτε, ο ηλεκτρονικός έλεγχος θα, γίνεται ε, μόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Τροπολογία 3, ε, Χάκιν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 9 καταπίπτει η 10 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται ε, το δεύτερο υπέρ κατά αποχές Πρέπει λοιπόν να κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα. Ε, ποιοι είναι παρακαλώ υπέρ αυτού του δεύτερου τμήματος. Ε, κατά έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Και αποχές. Πρόκειται για το δεύτερο τμήμα της 10. Έκλεισε η ψηφοφορία. 19 ε, κατά 18 υπέρ, το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ψηφίσουμε. Μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. Ε, πάμε τώρα στην τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Προφορική τροπολογία του κυρίου Μποστινάρου για τη 13. Θέλετε, μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Εγώ προτείνω να διαγράψουμε το EP Bodies γιατί σε οποιαδήποτε έκθεση μπορούμε να αναφερόμεθα μόνο σε επιτροπές του Κοινοβουλίου και σε βουλευτές δεν μπορούμε να αναφερόμεθα στη διοίκηση, στον Γενικό Γραμματέα και σε οποιοδήποτε άλλο διοικητικό στέλεχος. Αν λοιπόν γίνει αυτό αποδεκτό τότε και εγώ θα υπερψηφίσω. Ε, φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε με αυτό λέει ο Πρόεδρος με αυτή την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 14 όσοι έχει τροποποιηθεί υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παρακαλώ η τελική ε, ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Σας ευχαριστώ. Γκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, στην κυρία Σίνα. Τώρα θα περάσουμε στη ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Άουκεν. Αλλά πριν αρχίσουμε με την ψηφοφορία, νομίζω ότι δεχομένως υπάρχει μια αλλαγή στα αναπληρωματικά μέλη. Μα είπαν ότι η κυρία Σορνόσο αντικαθιστά τον Γιάννης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το έχουμε καταγράψει στον κατάλογο, έχει καταχωρηθεί και ως συνήθως θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Δεν θα ακολουθήσει μια συζήτηση, αλλά θα ακολουθήσει μια ψηφοφορία. Κυρία Όκεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, οι αναφέροντες ε, θα ψηφίσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερος ε, σημαντικό για πολλές χιλιάδες Ισπανούς ε, πολίτες και άλλους Ευρωπαίους πολίτες που επέλεξαν να ζήσουν στην Ισπανία ή σχεδιάζουν να εγκατασταθούν στην Ισπανία. Το σχέδιο ψηφίσματος δεν είναι κατά της Ισπανίας και θα ήθελα πραγματικά να το τονίσω. Επικρίνει ορισμένες πρακτικές που δυσχεραίνουν τη ζωή πολλών ανθρώπων και ζημιώνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το σεβασμό του περιβάλλοντος του ισπανικού πολιτισμού και της ισπανικής κοινωνίας. Αφορά την αρχή βάση της οποία, στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αφορά, ε, επικρίνει τη μαζική αστικοποίηση και τις επιπτώσεις της. Συγκρινόμενο με το αρχικό κείμενο και σαν αποτέλεσμα δύο πολύ επικοδοματικών συναντήσεων στο Στρασβούργο με τους ε, συναδέλφους, τους σκιώδης ηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες, από κοινού συμφωνήσαμε επί ενός αριθμού τροπολογιών που θεωρώ ότι επιφέρουν βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο, ε, το διευκρινίζουν, το καθιστούν περισσότερο ακριβές και αναδιατυπώνουν ορισμένες φράσεις και προσθέτουν κάποιες ε, κριτικές παρατηρήσεις. Ιδιαιτέρως άκουσα πολλά σχόλια και υποδείξεις των συναδέλφων καθώς και προτάσεις από μέλη όλων των πολιτικών ομάδων. Προσπάθησα να μεταχειριστώ με σεβασμό και κατανόηση πολλές ε, προτάσεις από τους Ισπανούς συναδέλφους που επίσης κατέθεσαν τροπολογίες, παρόλο που λυπούμε που δεν, είμαι σε θέση να, δεν, δεν σε θέση να αποδεχτώ πολλές από αυτές, γιατί στην περίπτωση αυτή θα καθιστούσαν το έγγραφο, ε, θα τοποθούν στο πλαίσιο μιας ενδοϊσπανικής διαμάχης και δεν θα ανταποκρινόντουσαν στα αιτήματα πολλών αναφερόντων, ε, οι οποίοι βλέπουν τις ζωές τους να επιδεινώνονται. Η, η τροπή καλείται να ασκήσει την ε, δημοκρατική της ε, κρίση επί των προτάσεών μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Άουκεν. Ε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα συμβαστικό κείμενο και όπως ξέρουμε συνήθως ψηφίζεται πρώτα το συμβαστικό κείμενο. Εκτός αν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις θα ήθελα να συνεχίσω και να σας παρακαλέσω να σκόσετε το χέρι και αν υπάρχει μια, ένα σχετικό αίτημα μέλους, μόνο τότε θα προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε, για να επιταχύνουμε και να αποφύγουμε τη σύγχυση. Γιατί να μην κινηθούμε όπως σε κάθε ψηφοφορία. Τώρα θα ψηφίσουμε τις παραγράφους 1 ως 5 που δεν υπάρχουν τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία, έχουμε το μέγιστο αριθμό των ψηφοφόρων. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής. 37 ψήφοι υπέρ, Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε τη λογική σκέψη A, α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 32 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Αυτό σημαίνει ότι η τροπολογία υπερθμονά είναι καταπίπτη. Ωραία, θα ψηφίσουμε την ενολογική σκέψη B. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 36 ψήφοι υπέρ. Μία αποχή. Τώρα, τροπολογία υπαρθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά. Ε, ζητήθηκε να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Έχει κανείς κάποια αντίρρηση από αυτού. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ Πρόεδρος, υποβλήθηκε ένα αίτημα και νομίζω ότι είναι σωστό. Εάν ένα μέλος θεωρεί ότι ενδεχομένως ε, ε, είναι, υπάρχει μια πλάνη, ένα σφάλμα εδώ, δικαιούται να ζητήσει ηλεκτρονική επαλήθευση. Όχι. Αποσύρθηκε. Επί ενός, κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό. Είμαστε εδώ για να ορίσουμε τις ε, απόψεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Νομίζω ότι κάποιος εδώ έκανε ένα σφάλμα εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, παρακαλώ να ελέγξετε. Οι άνθρωποι έχω την εντύπωση ότι φοβούνται τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές διαδικασίες. Κύριε ε, Μίτσελ, δεν μπορώ να ελέγξω μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ελέγξουμε I'm going to give the floor to the chairman of the committee. Ας δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής. Σύμφωνα με την άποψή μου, δεν υπάρχουν ε, ε, λόγοι για να επανεξετάσουμε το θέμα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, να μπορεί κάποιος να ψηφίσει και μετά να Υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ηλεκτρονικός ε, έλεγχος γίνεται μόνο εφόσον έχουμε ψηφίσει με ανάτες του χειρός και δεν είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν είμαι κατά του να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Ε, κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όσοι έχουν κάνει λάθος μπορούν να θέσουν το θέμα διαδικαστικά και εγώ ο ίδιος το έχω κάνει. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να ε, κάνουμε μία πρόταση για να λυθεί το θέμα είναι να ψηφίσουμε κατά πόσον θα πάμε πίσω και θα ελέγξουμε το αποτέλεσμα της ψηφορίας. Ε, στην περίπτωση αυτή θα συνεχίσουμε στην, για την επόμενη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα για τα εδάφια δέλτα έως... D2H που λέει. Εδάφια D2H. Κοιτάξτε, πρόκειται για την ψηφοφορία. Ε, πάμε τώρα στην ψηφοφορία για το D2H. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία, να ψηφίσουμε από τη μία την αιτιολογική σκέψη ΔΕΛΤΑΕΦ ε και μετά το GH από την άλλη. Μου είπαν ε, ότι για να ε, κατατεθεί έτοιμα για ξεχωριστή ψηφορία πρέπει αυτό να έχει κατατεθεί εκ των προτέρων. Δεν έγινε αυτό, γι' αυτό θα ψηφίσουμε ως έχει ο κατάλογος που μας έχει διανεμηθεί. Ψηφίσουμε τώρα για τα εδάφια D2H. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Ε, γκρίνεται 32 υπέρ, 2 h ψηφισατε ολοι εκλεισε η ψηφοφορια Πάμε στο recital, στο εδάφιο I. Ε, άρχεται η ψηφορία. Η τροπολογία νούμερο 3 είναι αυτή. Ψήφισετε όλοι, έκλεισε. Απορρίπτεται 21 ε, κατά, 14 υπέρ. Πάμε στην 4 με συμβαστικό ε, κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε 30 υπέρ, 4 κατά. Τροπολογία υπαριθμών 5. Είναι ψηφορία σε τμήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται 36 υπέρ. Τροπολογία υπαριθμών 6. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. «24 υπέρ, 11 κατά». Πάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 6. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Έκλεισε λοιπόν. Απορρίπτεται 15 υπέρ, 20 κατά. Ε, τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται 18 υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία υπαριθμών 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 8. Έκλεισε η ψηφοφορία. 23 κατά, 13 υπέρ, καταπίπτει. Τροπολογία υπαριθμών 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Μισό λεπτό. Ε, τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία για την 9. Έκλεισε. 25 κατά, απορρίπτεται τροπολογία 11 λεπρόδες, κάνει λάθος ε, σωστά με διορθώνονται λοιπόν. η 10 είναι έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται 25 υπέρ τροπολογία 12 άρχεται η ψηφοφορία έκλεισε εγκρίνεται 26 υπέρ η τροπολογία υπαριθμών 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται 26 περ Η 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 26 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε, απορρίπτεται 24 κατά. Τροπολογία υπεριθμών 15 ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε, εγκρίνεται 33 ε, υπέρ. Τροπολογία υπεριθμών 16, άρχεται η ψηφοφορία. Μισό λεπτό. Ε, ψηφίζουμε τώρα για την τροπολογία υπεριθμών 16. Ψηφίσατε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται 20 υπέρ. Τροπολογία υπεριθμών 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Απορρίπτεται 25 ε, κατά. Η 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Απορρίπτεται 22 ε, κατά. Η 19. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Ε, απορρίπτεται 23 κατά. Τροπολογία 20. Είναι ε, συμβαστικό κείμενο. Ε, άρχεται η ψηφορία. Μισό λεπτό. Ε, τροπολογία 20 λέει ο πρόεδρος. Τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. 21 είναι προσθήκη. Ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Τροπολογία υπεριθμών 22. Άρχεται η ψηφορία. Έκλεισε. 25 κατά. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία υπεριθμών 23. Άρχεται η ψηφορία. Έκλεισε. 26 υπέρ εγκρίνεται. Και κατόπιν τούτου νομίζω ότι η 24 καταπίπτει και πάμε στην 25 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε. Απορρίπτεται 27 κατά. Τροπολογία υπαριθμών 26. Άρχεται η ψηφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 19 επέρ 16 κατά. 27 ως εκ τούτου καταπίπτει και ψηφίζουμε για την 28 άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 24 ε, κατά. Ψηφίζουμε για την τροπολογία περιθμών 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε απορρίπτεται. 21 κατά. Η τροπολογία υπαριθμών 30 ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Είναι 31 ψήφισαν υπέρ. Τροπολογία υπαριθμών 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. εγκρίνεται 27 υπέρ, η τροπολογία αριθμών 32, άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται 30 κατά. Η 33 σε δύο τμήματα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Έκλεισε η ψηφοφορία. Κρίνεται 36, το δεύτερο τμήμα είναι μετά από εκεί που λέει δημόσιες κρατικές προμήθειες, άρχεται η ψηφορία, έκλεισε, ε, απορρίφθηκε 24 ε, κατά. Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 34. Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται 31 ψήφι κατά. Τροπολογία 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 26 ψήφους κατά. Και τώρα έχουμε την τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας απορρίπτεται με 26 ψήφους κατά. Τροπολογία υπαριθμών 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας τις ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 39. Ψήφισαν όλοι. Πέρας τις ψηφοφορίας Απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά. Τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 30 ψήφους κατά. Τροπολογία υπαριθμών 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία υπαριθμών 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά 43 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 32 ψήφοι υπέρ. Ο κύριος Μάιερ έχει μια προφορική τροπολογία για το δεύτερο τμήμα, αν δεν απατώμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι την απέστειλα εγκαίρως και λέει το εξή η προφορική τροπολογία. Υπάρχει μια νομοθεσία όπως στην περίπτωση της αρεγωνίας που υπάρχει μια αντιπαράθεση συμφερόντων μεταξύ πολιτών και τοπικών αρχών όσον αφορά την δημιουργία υποδομών σε αυτή την ζώνη. Υπάρχουν καθόλου αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Κυρία Άουκεν, έχετε αντίρρηση, είμαι υπέρ, λέει η κυρία Άουκεν. Και βεβαίω την έλαβα εγκαίρω, συνεπώ είναι δικό μου σφάλμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε ο κανονισμός λέει ότι αν υπάρχει μια αντίρρηση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την προφορική τροπολογία. Θα ψήσουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα χωρίς την προφορική τροπολογία. Ε, πρόκειται για την τροπολογία υπαριθμών 43. Ευχαριστώ κύριε Βίλαντ. Το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. Και τώρα θα περάσουμε στην ε, τροπολογία υπαριθμών 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες. 22 ψήφοι κατά. Τροπολογία υπαριθμών 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 29 ψήφους κατά. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας στις ψηφοφορίες απορρίπτεται 21 ψήφι κατά. Και τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία υπαριθμών 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας στις ψηφοφορίες απορρίπτεται με 26 ψήφους κατά. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίες ψηφοφορίες, απορρίπτεται 24 ψήφοι κατά. Τροπολογία υπερθμών 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 27 ψήφους κατά. Τροπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία Απορρίπτεται με 20 ψήφους κατά. 51. Συμβιβαστική τροπολογία. 51. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. απορρίπτεται με 19 ψήφους κατά. 52. Άρχεται η ψηφοφορία τώρα, λέει ο πρόεδρος, για την 52. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. Τροπολογία παριθμών 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 21 ψήφους κατά. Τροπολογία υπερθμών 54. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 20 ψήφους, 20 ψήφους κατά. 55. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 56 υπέρ 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. Η 57 καταπίπτει συνεπώς και περνάμε στην 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία υπαριθμών 60. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. 61. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά. 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ξέρω, τα λέω πολύ γρήγορα, υπερβολικά γρήγορα. Ε, απορρίπτεται 22 ψήφοι κατά. 63 άρχεται η ψηφοφορία. στις ψηφοφορίες εγκρίνεται 36 ψήφοι υπέρ. Η κυρία Σάντερ είναι εδώ. Θα πρέπει ένας από τους σοσιαλιστές να μην ψηφίσει. Η κυρία Σάντσεθ νομίζω αντικαθιστά... Σε κάποιος σας είχε ήδη αντικαταστήσει. Θα πρέπει να μας το πείτε. Όχι, η κυρία Σάντσο δεν θα ψηφίσει. Λοιπόν, ψηφίζουμε τις παραγράφους. Παράγραφος 1. Τροπολογία 64, άρχεται ψηφοφορία. ψηφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 26 ψήφοι κατά. 65, άρχεται ψηφοφορία. εγκρίνεται 35 ψήφοι υπέρ. 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 33 ψήφους κατά. 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας με 21 ψήφους υπέρ ε, εγκρίνεται. Διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χθε σας αποστήλαμε Αποστήλαμε στην κυρία Άουκεν, διαλογραφία, τη δυνατότητα ενό συμβασμού στον αφορά την παράγραφο 2 μεταξύ της τροπολογίας του κυρίου Πόπε και της δικής μας και επίσης την παράγραφο 3 με την ε, παράγραφο 64, 65, 66 και δεν λάβαμε καμία απάντηση. Δεν ξέρουμε αν, έχει, αν αποδέχθηκε τον συμβασμό ή όχι. Θα είχε ίσως την ευγενή καλοσύνη να μας απαντήσει η κυρία Άουκε. Δεν νομίζω ότι οι τροπολογίε αυτέ έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευση με την εισηγήτρια, αλλά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να δούμε κατά πόσο αυτέ οι συμβαστικέ τροπολογίε μπορούν να υιοθετηθούν η συγγήτρια. Δεν πρόκειται για συμβαστικέ τροπολογίες, δεν έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αντιβαίνουν στην έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Θα ψηφίσουμε σύμφωνα με τον κατάλογο ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε την 68. Άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. Ε, τροπολογία 69. Άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 28 ψήφους κατά. Ευχαριστούμε. Ε, η 70. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση στις εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. 71 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. 72 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση στις εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ. 73. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται με 21 ψήφου υπέρ. Η 74 έχει αποσυρθεί. Η 75 τώρα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι. Ε, μου είπατε ότι ε, το ε, έκλεισα υπερβολικά νωρίς. Ψηφίζουμε την 75. Ψήφισαν όλοι. Έκλεισε ψηφοφορία, απορρίπτεται με 21 ψήφους κατά και 14 ψήφους υπέρ. Η 76 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Έκλεισε ψηφοφορία. 70, ε, συγγνώμη, 28 ψήφοι υπέρ. Η 78 άρχεται η ψηφοφορία. 78. Μάλλον πρόκειται για την 77. Εδώ γράφει 78. Απορρίπτεται 27 ψήφοι κατά. Τώρα θα ψηφίσουμε την, ουσιαστική, την πραγματική 78. Άρχεται η ψηφοφορία για την 78. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφοι κατά, 12 υπέρ, απορρίπτεται. 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν νομίζετε ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μεταξύ της μιας και ψηφοφορίας και της άλλης, είναι επειδή έχουμε να κάνουμε ακριβώς με τεχνικά μέσα. Λοιπόν, 31 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, 29 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. Συνεπώς, Τροπολογία 81. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 ψήφοι πέρ 16 κατά. 82. Αρχη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 21 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται. 83. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 83. Όχι, λέει ο πρόεδρος. Μου είπαν ότι θα έπρεπε να έχει καταπέσει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε καταπέσει μόνο εφόσον η προηγούμενη τροπολογία είχε εγκριθεί. Καταπίπτει συνεπώς λέει ο πρόεδρος. Ωραία τότε θα περάσουμε στην επόμενη, την 85, εφόσον 84 καταπίπτει. 85, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες, απορρίπτεται με 24 ψήφους κατά. 86, άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα αρχίζει η ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος, για την 86. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 18 ψήφους κατά και 16 υπέρ. 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της απορρίπτεται με 20 ψήφους κατά. 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 20 ψήφους κατά. 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 25 ψήφους κατά. Η επόμενη, η 99 καταπίπτει και περνάμε στην 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 26 ψήφους κατά. Τώρα θα ψηφίσουμε την 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ. Ε, 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Εντάξει, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Περνάει με 22 ψήφους υπέρ. 97. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεν περνάει με 24 ψήφους κατά. 98. Αρχίζει η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Καταπίπτει με 27 ψήφους κατά. 98 το δεύτερο τμήμα. Αρχή η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 18 υπέρ. Το τρίτο τμήμα της 98. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Τώρα. Εγκρίνεται με 22 υπέρ. 98. Το τέταρτο τμήμα. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Η 99 καταπίπτει. Ψηφίσουμε την 100. Αρχής ψηφοφορία. Κύριε Πόπα, ζήτησα χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα είναι μέχρι το παράκτιο περιβάλλον, coastal environment. Συμπεριλαμβάνει και τις λέξεις coastal environment. Όχι. Χωριστή ψηφοφορία. Ναι, λέει ο πρόεδρος, το κατάλαβα αυτό. Αλλά πού θα γίνει ο διαχωρισμός. Το δεύτερο τμήμα αρχίζει στο Coastal Law, ο νόμος για τις παράκτιες περιοχές. Έτσι. Αυτό είχα πει στην αρχή και δεν έγινε αποδεκτό. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το δίκαιο για τις παράκτιες περιοχές, to revise the coastal law. Υπάρχει αντίρρηση για τη χωριστή ψηφοφορία, κύριε Πόπα. Κύριε Άουκεν, κύριε Πρόεδρος, για να είμαστε δίκαιοι, διακόπτεται ο Πρόεδρος. Κάντε μια χειρονομία καλή θέληση, κύριε Άουκεν, ε, να γίνει δηλαδή αυτή η χωριστή ψηφοφορία. Να σας διαβάσω μέχρι το τέλος του πρώτου τμήματος αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ισπανικών αρχών να προστατεύσουν το παράκτιο περιβάλλον και όπου είναι δυνατόν να ανακτήσουν το παράκτιο περιβάλλον. Αυτό είναι το, πρώτο, το τέλος του πρώτου τμήματος. Εντάξει κύριε Ποπα, ναι. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα. Αυτό είναι η τροπολογία 100. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Είναι αυτό που θέλατε, έτσι. Τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα. Έχετε καταλάβει ποιο είναι. Ναι. Ψηφίσαν όλοι. Το δεύτερο τμήμα πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Πάμε στην 101. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ και 12 κατά. 102. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 27 ψήφους κατά. 103. Τροπολογία 103 του κυρίου Πόπα. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ. Η επόμενη καταπίπτει και ψηφίζουμε τώρα την 106 γιατί καταπίπτει και 105. Πάμε στην 106. Έτσι, ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται με 31 ψήφου υπέρ. Τροπολογία 107. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία απορρίπτεται με 20 ψήφους κατά. 108. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται με 20 ψήφου κατά. 109 αυτή καταπίπτει. 110 ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Μου λέτε ότι απο... έχει αποσυρθεί εγώ δεν το είχα στον κατάλογό μου, αλλά νομίζω θα καταψηφιστεί που είναι σαν να έχει καταπέσει. Δεν ασχολούμαστε λοιπόν άλλο. Πάμε στην 111. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 20 ψήφους κατά. 112 καταπίπτει. 113 ή Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται με 27 ψήφους. Κατά. 114. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται με 31 ψήφους. Κατά. 115. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 18 κατά, 17 υπέρ απορρίπτεται. 116. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. 117. Ψηφοφορία τώρα. Πέρας ψηφοφορίες. 31 ψηφοί υπέρ. Γκρίνεται. 18, 118. Αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ. 119 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 21 ψήφους κατά. 20 Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται με 21 ψήφους κατά. 121. Αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. 122 της κυρίας Όκεν. Αρχή ψηφοφορία. Ψηφίσατε. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. 123. Ψηφίζουμε την 123. Πέρας. Ε, δεν περνάει με 23 ψήφους κατά. 124. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. Ψηφίζουμε την 125. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 27 ψήφους κατά. 126. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 29 ψήφους κατά. Πάμε στο 127. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας φοφορίας απορρίπτεται με 29 ψήφους κατά. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος όπω τροποποιήθηκε. Αρχή ψηφοφορία παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Μιλήσα τώρα ποτέ κύριε Μίτσελ. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ και 11 ψήφους κατά. Μία αποχή. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Αλλά συγχαρητήρια και στην Επιτροπή για τον παραδειγματικό τρόπο με τον οποίο αυτή η μακρά και κουραστική ψηφοφορία διεξάγει. Και τώρα ξανά στον πρόεδρο. Ο κύριος Μίτσελ, πρέπει να σας ανακοινώσω κάτι για τον κύριο Μίτσελ, παρακαλώ. Ο κύριος Μίτσελ έβγαλε την κάρτα του ε, νωρίτερα. Ε, άρα έχουμε μία ψήφο επιπλέον υπέρ. 24 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια κυρία Όκεν για τη θαυμάσια έκθεση αυτή. Πρόεδρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάικλ Κάσμαν που ήταν πρόεδρος, προείδρευσε σε αυτή τη δύσκολη ψηφοφορία. Ξεπέρασε όλα τα εμπόδια που του βάλαμε με παραδειγματικό τρόπο. Θα δώσω το λόγο, αν επιτρέπετε, στην κυρία Άουκεν, πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο για μία δύσκολη. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή πολύ θερμά για την υποστήριξή της σε αυτή τη τόσο δύσκολη έκθεση. Ήταν σαφές ότι εδώ πρόκειται για, για συγκεκριμένα συμφέροντα και βεβαίως ε, υπήρχαν και επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο. Και από την άλλη ήταν πολύ θετικό που μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι υπήρξαν και Ισπανοί συνάδελφοι οι οποίοι υποστήριξαν την έκθεση αυτή. Γιατί πρόκειται βεβαίω για την κατάσταση στην Ισπανία αλλά και για την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και πραγματικά τέθηκε η έκθεση στο επίπεδο που τη αρμόζει γιατί πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντο και για την προστασία του πολιτισμού. Και Ελπίζω η Κομισιόν πραγματικά να ακολουθήσει αυτές τις πολύ ξεκάθαρες υποδείξεις μας. Σας παρακαλώ, βγάλτε τις ε, κάρτες σας από το μηχάνημα. Ας δώσω το λόγο στον Πρόεδρο για να πάμε στο επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ όλους τους συντονιστές, τους κοιόδης εισηγητές που ασχολήθηκαν με αυτή τη μακρά ψηφοφορία. Μακρά και δύσκολη. Please sit down and take your place. Καθίστε παρακαλώ και να ξεκινήσουμε. Ε, ευχαριστώ εκ νέου τον Μάικλ Κάσμαν που προείδρευσε αυτή τη δύσκολη ψηφοφορία. Έχει μεγάλη ικανότητα σε αυτό. Προχωράμε λοιπόν τώρα, κυρίε και κύριοι. Το σημείο 23 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για μια έκθεση από την διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία. Είναι το σημείο 23 και έχετε το έγγραφο. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι οι λίγες τροπολογίες που υποβλήθηκαν από την κυρία Στροκόβα έχουν γίνει αποδεκτές. Τις έχω μπροστά μου. Φαντάζομαι λοιπόν ότι έχουν γίνει αποδεκτές. Υπάρχει πρόβλημα. Γιατί κουνάει το κεφάλι σας, Πρόεδρε. Όχι, δεν έχουν γίνει δεκτές οι τροπολογίες. Αλλά θα φτάσω μια στιγμή και σε αυτό. Ναι, ξέρω για ποιες μιλάτε. Θα μιλήσω και για τις τροπολογίες. Σιγά σιγά. Το κάθε πράγμα στον καιρό του. Έχετε το έγγραφο αυτό μπροστά σας, κυρίες και κύριοι. Τα μέλη της αποστολής ε, στην Βουλγαρία ήταν ο Μάρτιν Λεμπίσκι, η κυρία Σίνοτ και ο Ντέιβιτ Χάμερστάιν Μίντς. κυρία Στροκόβκα ήταν ένα μέλος αποστολής εξοφίσιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα μέλη της Επιτροπής μας δεν μπορούν να είναι επίσημα μέλη μιας αποστολής που γίνεται στη χώρα τους. Η κυρία Στροκόφα ήταν μαζί μας, την ευχαριστώ που ήταν μαζί μας, αλλά δεν ήταν μέλος αυτό καθεαυτό της ε, αποστολής στη Βουλγαρία. Δεν θέλω να σπαταλάω χρόνο τώρα, δεν θα επαναλάβω το περιεχόμενο του εγγράφου. Το έχετε τους φακέλους σας. Και αν ένα από κάποιο από τα μέλη της αποστολής που πήγαν στη Βουλγαρία θέλουν να πάρουν το λόγο, κυρία Σίνο, το κύριος Χάμερστάιν Μίντς, ε, μπορούν να πάρουν το λόγο. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Εν συνεχεία θα σχολιάσουμε μόνο τις τροπολογίες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν ε, συμμετείχα σε αυτή την αντιπροσωπεία. Θέλω όμως να πω κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Ίσως εγώ δεν κατάλαβα καλά. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξής. Αν κατάλαβα καλά, τα μέλη της ε, χώρας, από την χώρα την οποία επισκεπτόμεθα, είναι εξοφίσιο ε, μέλη της ε, αντιπροσωπείας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο και να μην αγνοούνται. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι όταν οι αντιπροσωπείες επισκέπτονται μια χώρα δεν ε, μπορούν όλα τα εξοφίσιο μέλη να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις και δεν αντιμετωπίζονται ως μέλη κανονικά της αντιπροσωπίες, Ενώ το αντίθετο θα πρέπει να ισχύει. Ακριβώς επειδή εξοφίσιο είναι μέλη της αντιπροσωπείας, αυτόματα αποτελούν ε, μέλη της αντιπροσωπείας αυτή, θα έπρεπε να τους αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο πρόεδρος. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για παρεξήγηση εξ officio. Στην περίπτωση αυτή δεν σημαίνει ότι αυτόματα συνυπολογίζονται στην αντιπροσωπεία. Το αντίθετο είναι εκτός αντιπροσωπείας. Τώρα κατά πόσον αυτό είναι παραπλανητικό ή όχι δεν το γνωρίζω. Όταν λοιπόν ε, πήγαμε στην Πολωνία, εγώ παραδείγματο χάρη δεν συμμετείχα σε κάποιες ε, συζητήσεις ε, που έγιναν σε ένα Υπουργείο γιατί ο κύριος Χάμερσταϊν Μίντς είχε αντιρρήσεις. Ήθελα να επισκεφθώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τότε ο κύριος Χαμαστάιν ε, Μίντς ε, είπε ότι δεν γίνεται αυτό γιατί δεν ήμουν κανονικά μέλος της ε, αντιπροσωπείας. Το δέχθηκα λοιπόν και η πεπατημένη αυτή είναι δεν μπορεί κανείς να συνυπολογίζεται σε μία αντιπροσωπεία όταν ε, μία αντιπροσωπεία επισκέπτεται τη χώρα του βουλευτή. Εγώ ε, διαφωνώ κάθετα με αυτό που λέτε εσείς ως ερμηνεία ε, του τι είναι μέλος εξοφίσιο. Αυτό σημαίνει ότι είστε αυτόματα μέλος μιας αντιπροσωπείας και όταν η αντιπροσωπεία επισκέπτεται τη χώρα σου τότε έχεις να παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο και όχι το αντίθετο που λέτε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πιστεύω ότι εδώ ε, ακολουθούμε λάθος κατεύθυνση. Πρόεδρε, δεν μ' αρέσει που παρεμβαίνω ανάμεσα σε δύο δικηγόρους, αλλά ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι ο συνάδελφος έχει δίκιο. Εγώ, όπως ε, ερμηνεύω τον όρο εξοφίσιο, αυτό σημαίνει ότι συμμετέχει κανείς ε, σε οτιδήποτε διαδραματίζεται. Εντάξει, δεν μπορεί κανεί να ψηφίσει, μπορεί όμω ε, κάλλιστα να εμφανίζεται κανεί. Εγώ, παραδείγματο χάρη, είμαι εξοφίσιο, μέλο ε, του ε, Προεδρείου των Βρετανών Συντηρητικών και εμφανίζομαι σε κάθε συνάντηση. Το άλλο το βρίσκω γελίο. Ε, Ένα άνθρωπο που ξέρει εξορισμού πράγματα για τη χώρα, όπω εσεί στην Πολωνία ή η κυρία Στάκοβα, ε, το να εμποδίζεται να συμμετέχει, αυτό είναι τρελό. Το να μην μπορεί να ψηφίζει, εντάξει, με αυτό συμφωνώ, αλλά το να συμμετέχει στην επιτροπή, αυτό είναι αυτονόητο. Ε, και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ερμηνεία και όχι αυτό που λέτε εσείς, γιατί αυτό που λέτε εσείς φοβάμαι ότι είναι λάθος. Πρόεδρος, εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα πριν από πάρα πολλά χρόνια όταν ε, συστήθηκε η Επιτροπή ή στην αρχή αυτής της θητείας. Από τότε που έγινα εγώ μέλος της Επιτροπής δέχθηκα ότι ισχύει αυτή η ερμηνεία που σας παρουσίασα. Τώρα, αν ο Sir Robert Atkins εργάζεται ε, στον κώδικα best practice ε, για την Επιτροπή μας, ε, τότε είναι προφανές ε, ότι θα πρέπει να πει και την άποψή του. Αυτή η επιχειρηματολογία είναι αποδεκτή. Δεν είναι όμως ε, δυνατόν η άποψη ενός μέλους της Επιτροπής η οποία επισκέπτεται μια χώρα να αγνοείται. Το αντίθετο, εγώ θα ήθελα ευθύς εξ αρχής την κυρία Στάρκοβα να, δώσετε, να τους δώσετε το λόγο και πριν από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Δεν είναι δηλαδή αλήθεια ότι αγνοούμε τις απόψεις που εκφράζονται από αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτή όμως είναι μια συζήτηση η οποία έτσι και αλλιώς εξορισμού είναι ξεπερασμένη. Κυρία Σίνετ, κοιτάξτε, σχετικά με το θέμα το εξοφίσιο, και κοιτάζοντας λίγο την ε, fact-finding ε, αποστολή που πήγε στην Ιρλανδία, τα εξοφίσιο μέλη είναι πολύ καλό που συμμετέχουν σε μια αντιπροσωπεία γιατί γνωρίζουν καλά τα τοπικά γεγονότα. Αλλά αν πάμε στην περίπτωση της Ιρλανδίας, εκεί έχουμε περισσότερους ε, Ιρλανδούς από ό,τι ήταν τα μέλη της αντιπροσωπείας. Και ο λόγος που τα μέλη, τα εξοφίσιο πρέπει να απομονώνονται είναι γιατί ε, θα πρέπει να εισακουστούν οι απόψεις των εθνικών ε, βουλευτών. Είναι λοιπόν ε, μια fact-finding mission και είναι σημαντικό να υπάρχει αντικειμενικότητα. Εγώ συμμετείχα σε αυτήν την επιτροπή για την Ιρλανδία, αλλά ήξερα πάρα πολύ καλά ότι για να υπάρχει αντικειμενικότητα, ήξερα βέβαια πολύ καλά το τι γίνεται, αλλά ήταν πολύ σωστό το ότι δεν συμμετείχα στην αντιπροσωπεία. Γιατί όλοι οι Ιρλανδοί που ήμασταν ξεχωριστοί από την αντιπροσωπεία ε, ακριβώ λόγω του ότι εμπλέκεται και η εθνική πολιτική. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ε, ε, πολύ σημαντική ερμηνεία. Ακόμα και αν εμένα δεν με βόλευε στην Ιρλανδία, ο κανόνας ε, παραμένει και είναι σημαντικός. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα επ' αυτού. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ λοιπόν ε, προτείνω τώρα να μπούμε στην ουσία του θέματος, Sir Robert Atkins. Ε, κοιτάξτε, αναφέρεται εκεί ότι οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εκφράσει απόψη του στην αρμόδια επιτροπή. Η κυρία Στάρκοβα έχει καταθέσει τροπολογίες και ως εκ τούτου πρέπει να εισακουστεί η άποψή της. Sir Robert, Ανακοίνωσα όμως ότι ε, θα εκφραστούν οι απόψεις της και τώρα θα έλεγα να μπούμε στην ουσία διαδικαστικό αυτό που θέλετε να πείτε. Βεβαίως, εντάξει, πέστε το διαδικαστικό αν θέλετε. Όταν εγώ ήμουνα σε μία αποστολή fact-finding όπως αποκαλείται, ε, ε, συντάξαμε ένα έγγραφο για την αποστολή αυτή. Το έγγραφο αυτό αποκαλύφθηκε έγγραφο εργασίας και δεν τροποποιήθηκε. Ε, όταν συντάξαμε το έγγραφο τότε λάβαμε υπόψη της ε, λάβαμε υπόψη της απόψης όλων των Ιταλών γιατί η Επιτροπή αυτή πήγε στην Τοσκάνα. Ήταν λοιπόν ένα έγγραφο εργασία και δεν τροποποιήθηκε. Ε, μπορείτε αν θέλετε να ακούσουμε όσε τροπολογίε θέλετε, αλλά δεν τροποποιούν αυτέ το κείμενο. Πρόεδρος, ο κύριος ε, Ντεμέτερ, αν άκουσα καλά το από την Επιτροπή παρακαλώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τώρα τι να πω, δεν, δεν έχω τίποτα να πω. Λυπάμαι. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ε, πρόεδρος, τότε ε, κερδίσαμε κάποιο χρόνο. Κυρία Στάρκοβα, κοιτάξτε, ε, εγώ θέλησα να καταθέσω αυτές τις τροπολογίες για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στις ε, συστάσεις προς την κυβέρνηση. Γιατί είχαμε πολλές συναντήσεις και ακούσαμε πάρα πολλού αναφέροντες. Ε, τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη Βουλγαρία διαφέρουν. Εγώ λοιπόν αυτό ακριβώς σκέφτηκα, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι και γι' αυτό το λόγο διένυμα τις τροπολογίες αυτές στους συναδέλφους μου που είναι κανονικά μέλη της αντιπροσωπείας και όχι εξοφίσιο μέλη. Εφόσον λοιπόν οι συνάδελφοι στηρίζουν τις τροπολογίες μου, ε, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνουν αποδεκτές. Παρότι ε, συμφωνώ μαζί σας αν θέλετε ότι είμαι μέλος εξοφίσιο στην ε, Επιτροπή αυτή. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ε, επικοδομητική σας στάση. έχετε μπροστά σας το κείμενο της κυρίας Στράσκοβα ε, όσον αφορά το σημείο υπαριθμών 1, συμφωνώ, δεκτό, ε, σημείο υπαριθμών 2, δεν γνωρίζω γιατί απορρίπτουμε ή πρέπει να απορρίψουμε την έκκληση αυτή προς την βουλγαρική κυβέρνηση. Η κυρία Στάρκοβα είναι υπέρ του να διαγραφεί, εγώ θέλω να παραμείνει. Όσον αφορά την τροπολογία όπου καλούμε την ε, βουλγαρική κυβέρνηση ε, να προβεί σε αξιολόγηση, συμφωνώ με αυτό. Και κατόπιν όσον αφορά την αναφορά, νομίζω ότι είναι πιο λογικό να έχουμε μια γενικότερη διατύπωση, γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι εμείς προτιμούμε κάποιες αναφορές έναντι κάποιων άλλων. Όσον αφορά λοιπόν τι ε, τροπολογίε ε, της κυρίας Στράκοβα, ε, πρώτη πέρ κατά τις δύο, υπέρ της τρία κατά της τέσσερα. Και εάν κάποιος άλλος θέλει το λόγο, παρακαλώ, αλλιώς θα ρωτήσω την κυρία Στράσκοβα κατά πόσον συμφωνεί. Sir Robert Atkins. Εγώ δεν νομίζω ότι οι δύο πρέπει να διαγραφεί υπάρχουν άλλες τροπολογίες που τη στηρίζουν. Καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Στράσκοβα, αλλά εάν ε, διαγραφεί αυτή όπως λέει και ο πρόεδρος και προσθέσετε κατόπιν της άλλης τροπολογίες εγώ νομίζω ότι ενισχύεται το κείμενο και δεν αποδυναμώνεται ε, κατόπιν να ορίσουμε τις ε, δυνατότητες αποζημίωσης αυτό είναι ναρκοπαίδιο θα έλεγα και αν δεν συμφωνήσουμε στην Επιτροπή για μία διατύπωση η οποία ε, θα είναι λιγότερο ε, επιβλητική, ε, εντάξει, θα μπορούσαμε να τα αποσύρουμε. Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε να προτείνετε η Επιτροπή Αναφορών θα εξετάσει το συντομότερο δυνατόν τα θέματα αυτά. Ε, κοιτάξτε, αυτό, με αυτό εγώ αν θέλετε συμφωνώ και αν βοηθάει και τους ε, αναφέροντες ε, να το δούμε το συντομότερο των τον Δεν, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν πρόεδρε ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε κυρίως ε, όσον αφορά αυτό το θέμα της αποζημίωσης που όπως σας είπα είναι πολύ λεπτό το θέμα. Κατά τα άλλα η ε, συνάδελφος Σάσκοβα προτείνει πολύ σωστά πράγματα και πρέπει να δεχθούμε αυτά που προτείνει με οποιαδήποτε ιδιότητα κρίνουμε ότι καταθέτει τις τροπολογίες της. Πρόεδρος, Κατόπιν τούτου επαναλαμβάνω. Τροπολογία υπαριθμών 1. Εγκρίνεται. Εδώ έχουμε μία ε, παρένεση προς την Κομισιόν να δρομολογήσει έρευνες. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα από αυτού. Συμφωνείτε να παραμείνουμε, να δεχθούμε αυτή την πρόταση που λέει ότι απευθύνουμε έκκληση προς την βουλγαρική κυβέρνηση. Βεβαίως ο κύριος Χάμαστάν Μίντσε και άλλα μέλη της Επιτροπής δεν είναι παρόντα. Ερωτώ, εσείς είστε υπέρ αυτής της παρένεσης προς την κυβέρνηση. Ωραία. Τρία. Και για αυτήν είμαι υπέρ. Και το τελευταίο σημείο βρίσκεται στην τελευταία σελίδα. Συμφωνείτε με αυτό. Δηλαδή την ε, αναφορά να μην την αντικαταστήσουμε γιατί αυτό θα προκαλούσε την εντύπωση ότι κάποιες άλλες ε, τις ε, αγνοούμε. Πρόεδρε, το θέμα είναι ότι είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις και ορισμένες ε, αναφορές κατ' ουσίαν δεν είναι αναφορές, δηλαδή δεν έχουν καταχωρηθεί επίσημα. Το να παραμείνουμε γενικοί στη διατύπωση, αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνουμε στην έκθεση και τους ε, αναφερόμενους εισαγωγικά, που δεν είναι ακριβώς αναφερόμενοι γιατί δεν έχουν καν αριθμό καταχώρησης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, είχαμε πάρα πολλές άτυπες συναντήσεις με πολλούς ε, ιονοί αναφερόμενους, ε, που εντάξει είναι κατά κάποιον τρόπο αναφερόμενοι, αλλά δεν έχουν στείλει ακόμα την αναφορά τους ε, στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Πρόεδρος, μα ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή τη γενική διατύπωση που περιέχει το κείμενο και δεν θα ήθελα να είμαι πιο συγκεκριμένος νομίζω και ο Sir ε, Robert ε, συμφωνεί ε, να παραμείνουμε σε αυτούς τους αναφερόμενους που είναι επίσημα καταχωρημένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, Νομίζω ένα σημαντικό πράγμα σε αυτήν την Επιτροπή είναι ότι η Επιτροπή έχει μια τάση να περικλεί και όχι να αποκλείει πράγματα. Και ένα πράγμα που έχει σημασία με μια αποστολή επιτόπια fact-funding είναι ότι οι άνθρωποι έρχονται και βλέπουν την Επιτροπή και αυτό δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Ε, χρησιμοποιώντας τον όρο ε, αναφορά, εντάξει... Ε, υπάρχει κάποια ερμηνεία το τι ακριβώς σημαίνει. Ας το πούμε κάπως γενικότερα. Όταν πάμε σε μια χώρα, οι άνθρωποι έρχονται εκεί με τις αναφορές τους, με τα αιτήματά τους, αν θέλετε. Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Σίνοτ ε, συμμετείχε στην ε, αντιπροσωπεία, το ίδιο και ο υποφαινόμενος και για τους ε, λόγους που αναφέρθηκαν ε, θα έλεγα να παραμείνουμε στη γενική διατύπωση. Ο κύριος Χάμεσταν Μίντς ε, δεν είναι παρόν, λέει ο πρόεδρος. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ψηφίσουμε. Κοιτάξτε, σε Robert λέει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Και στην Βουλγαρία το ίδιο ισχύει. Συμφωνώ με την Κάθη ότι πράγματι Κάποια από αυτά τα αιτήματα δεν είναι επίσημες αναφορές, μπορεί να είναι ε, δυσαρέσκεια, ανησυχία. Ε, πράγματι πρέπει να είμαστε ε, πολύ προσεκτικοί πώς θα ρυθμίσουμε το θέμα. Γιατί εφόσον δεν υπάρχει επίσημη καταχώρηση δεν ξέρουμε και πώς είναι αυτά τα αιτήματα. Ίσως μπορούμε να βρούμε κάποια διατύπωση πριν τελειώσει η συνεδρίαση που να είναι ευρέως αποδεκτή και θα βοηθήσει αυτή η διατύπωση τους ενδιαφερόμενους να εκφράζουν την ανησυχία τους και παράλληλα ε, δεν ε, θα ε, δημιουργείται πρόβλημα. Πρόεδρος. Έχω την εξής πρόταση να κάνω. Ε, συμφωνείτε οι αιτήσει που έχουν καταχωρηθεί και άλλες, να συμπεριλαμβάνει το κείμενο τις επίσημες καταχωρήσεις και άλλες με τις οποίες έχουμε εμπλακεί, τις οποίες έχουμε εξετάσει κατά κάποιον τρόπο. Πολύ ωραία. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη εγκρίνουμε αυτήν την ε, έκθεση και το επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας ε, διάταξης είναι το 24 24. Όχι, το 25. Ο κύριος ε, Τομπίας Μπίεμαν, εξ ονόματος της ε, Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στην αναφορά 0828 του 2006. Ε, πρόκειται σε αυτή την αναφορά. Ο αναφέρον λέει ότι δεν ζητήθηκε γνώμη του πριν ε, από το χαρακτηρισμό ζωνών ασφαλείας στο αεροδρόμιο. Στην ε, συνδύαση επιτροπή Επιτροπής το περασμένο Ιούνιο, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε από τον αναφέροντα να παράσει περισσότερες πληροφορίες. Σε μία επιπλέον επιστολή της 23 Σεπτεμβρίου του 2008, ο αναφέρον επαναλαμβάνει ότι ε, διαπίστωσε παραβίαση της οδηγίας σε σχέση με την ευθύνη της Επιτροπής όσον αφορά ε, αυτές τις ζώνες ασφαλείας ή ελέγχου στα αεροδρόμια. Ο αναφέρον αναφέρεται ε, στις ε, διατάξεις ε, σχετικά με τις ε, περιοχές σε Βέζο. Ο στόχος αυτών των διατάξεων αφορούν τις σωστές αποστάσεις μεταξύ χημικών βιομηχανιών. σε σχέση με κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν δύο λόγια τους οποίους η οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε σχέση με αυτή την αναφορά. Οι διατάξεις ε, στην οδηγία αφορούν την κατασκευή νέων βιομηχανικών χημικών εγκαταστάσεων ή τις, ε, ανάπτυξη γύρω από αυτά τα εργοστάσια. Ε, και στην περίπτωση αυτή προποθέτει μια διαβούλευση με το κοινό. Αλλά στην περίπτωση που περιγράφει ο αναφέρον, η οδηγία αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν υπήρξαν νέα ε, βιομηχανικά, χημικά ε, εργοστάσια στην, εποχή, στην περιοχή αυτή και όσον αφορά τα υπάρχοντα εργοστάσια δεν εμπίπτουν σε τάξεις οδηγίας. Κατά δεύτερο λόγο, η οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί, από τις, να μεταφερθεί στη χώρα τώρα μέλος το 99 αλλά ο αναφέρον αναφέρεται στις ζώνες ασφαλείας στα αεροδρόμια το 1993 και την εποχή εκείνη η οδηγία αυτή δεν είχε τεθεί σε ισχύ και επομένως δεν ήταν εφαρμοστέα. Επιπρόσθετα ο αναφέρον επίσης ε, δηλώνει παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων στον τόπο εργασία τους. Αυτή η οδηγία αναφέρεται στις ε, προϋποθέσεις, στην υποχρέωση των εργοδοτών να ε, εξασφαλίσουν σωστές ε, συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους. Εν κατακλείδη, θέλουμε να πούμε ότι λυπούμεθα για τον αναφέροντα, αλλά στη βάση των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μπόρεσε ε, δεν μπόρεσε να αποδεχθεί καμία παραβίαση των οδηγιών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ έχουμε παρόντα τον αναφέροντα, τον κύριο Κίλιγκαν. τον εκπρόσωπό του μάλλον του κυρίου Κίλιγκαν, ε, ο οποίος έχει το λόγο. Uh, Mr. Um, Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ τον κύριο Γκέλιγκαν, ο οποίο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ και θα ήθελα να εκπροσωπήσω την υπόθεσή του. Άκουσα να φέρει συζήτηση προηγουμένω η έννοια δημοκρατία. Ε, δεν νομίζω ότι αναφέρεται εδώ, ε, ότι εφαρμόζεται εδώ σχέση με αυτή την ε, οδηγία. Και δεν διαβολεύτηκαν καθόλου οι ιδιοκτήτες της γης, καθώς και οι πολίτες οι οποίοι πλήττονται από αυτά τα μέτρα. Δεν υπήρξε καμία δημοσίευση στον τύπο σε σχέση με τις προθέσεις του κράτους να χαρακτηρίσει αυτές τις ζώνες ασφαλείας. Δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση αυτών των ζωνών, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δεν έγινε καμία επιστημονική αξιολόγηση και δεν ζητήθηκε η γνώμη τρίτων μελών, μερών, όπως ε, προβλέπει η οδηγία. Δεν δόθηκαν επίσης καθόλου λεπτομέρειες όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου. Το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας στην Ιρλανδία είναι εντελώς ε, δυσανάλογη ενώ κανονικά θα πρέπει να βασίζονται οι ορισμοί αυτοί σε επιστημονικές αξιολογήσεις των κινδύνων. Υπάρχουν 92 τέτοιες ζώνες στην Ιρλανδία χωρίς να έχουν γίνει αυτές οι σωστές αξιολογήσεις κινδύνου. Όλο το πρόγραμμα αυτό στερείται διαφάνειας ε, νομίζω θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ρύθμιση. Υπάρχει μια ολόκληρη κίνηση στην Ευρώπη προς την κατεύθυνση μιας σωστότερης ρύθμισης. Ε, πρόκειται για μια παραβίαση εδώ και της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών. Επίσης δεν είναι συμβατό το πρόγραμμα αυτό με την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. ε, στη, υπάρχει Κατετέθηκε λοιπόν ε, μια ε, προσφυγή γιατί ο άνθρωπος αυτός ε, δεν είχε καμία ιδέα για το πώς χαρακτηρίστηκε η περιοχή και δαπάνησε και πολλά άλλα χρήματα ε, ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπάρχει ένα πρόσκομα και κύριε Πρόεδρε η κατάσταση είναι η εξής ότι η ΡΑΣ και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτές τις ζώνες Σέβεζο πράγματι έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα διότι σε αυτό το εργοστάσιο αποδίδεται μία έκταση η οποία δεν είναι σε συμφωνία με την ε, προηγούμενη οδηγία. Είναι η περίπτωση όπου οι ζώνες αυτές στο Σέβεζο ανήκαν ακριβώς στην εταιρεία στο εργοστάσιο ΡΑΣ. Εγώ θέλω να πω εξ ονόματος του αναφέροντος ότι αυτές οι οδηγίες έχουν σχέση με την ασφάλεια. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Προφανώς και στηρίζουμε την ασφάλεια που προβλέπεται αυτή η οδηγία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την οδηγία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την Ευρώπη. Προφανώς και είμαστε υπέρ της ασφάλειας, αλλά διαφωνούμε αυτή η οδηγία να εφαρμόζεται εργάζεται αποκλειστικά και μόνο στην Ιρλανδία. Και γι' αυτό θα θέλαμε να ερευνήσετε περαιτέρω το θέμα, να υπάρχει σωστή εφαρμογή. Εξάλλου, ε, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο όσοι κάνουν ανάλυση κινδύνου επιτόπου να κάνουν σωστή ανάλυση του κινδύνου και να μεταφέρουν το περιεχόμενο αυτής της ανάλυσης ως ενημέρωση σε όλους τους πολίτες. Στην Ιρλανδία εδώ και χρόνια αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει σωστά και έτσι λοιπόν τα εθνικά, το εθνικά αεροδρόμια και τα τοπικά έχουν αρνηθεί σε πολίτες να εκμεταλλευτούν την ιδιοκτησία τους. Ε, το καλοκαίρι βρήκαμε ότι προτείνεται ε, να χτιστεί μια νέα ε, πόλη σε αυτή την ίδια περιοχή που υποτίθεται αμφισβητείται και μάλιστα και πολυόρφα κτίρια. Αλλά βλέπετε ότι εδώ εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχω και μία σύντομη περίληψη της αναφοράς. Αν θέλετε μπορώ να στείλω την αναφορά αυτή σε όλα τα μέλη. Σας λέω, επαναλαμβάνω, δύο μέτρα και δύο σταθμά εφαρμόζονται κυρίως όσον αφορά αυτή την οδηγία και υπάρχει και πλήρης έλλειψη διαφάνεια για να ξέρουμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται αυτές οι ε, οδηγίες περί ζωνών Σέβεζο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, καμία διαφάνεια και σε έλλειψη λογοδοσίας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω τον αναφέροντα. Είμαι μέλος του Κοινοβουλίου. Σε αυτή την περιοχή. Σε αυτή την περιοχή στην οποία αναφέρεται ο αναφέρον. Και ο βασικός λόγος αυτής της αναφοράς είναι ο τρόπος με τον οποίο η ζώνη αυτή χαρακτηρίστηκε ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίστηκε δεν ε, κοινοποιήθηκε στους ανθρώπους που πλήττονται από την απόφαση αυτή. Υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή παραβίαση. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος γιατί σας έφτασε εδώ αυτή η αναφορά. Δεν αμφισβητούμε την εμβέλεια της ε, οδηγίας. Δεν υπάρχει καμία ε, διαφάνεια απέναντι στους ιδιοκτήτες. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνήσουμε. Ότι δεν ενημερώθηκαν δηλαδή οι ιδιοκτήτες. Γιατί Υπάρχει ένα σοβαρό το πρόβλημα εδώ σε ό,τι αφορά τον τρόπο μεταφοράς της, της οδηγίας στην Ιρλανδική νομοθεσία. Και κάτι άλλο. Το θέμα αυτό επηρεάζει τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την αντιλαμβάνεται ο κόσμος ως έναν οργανισμό ο οποίος επιβάλλει νόμους εκ των άνω στους ανθρώπους, χωρίς κοινοποίησεις, χωρίς ενημέρωση μέσω των εφημερίδων κτλ. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω τον κύριο Γκίλγκεν, τον αναφέροντα, και να σας ζητήσω, Πρόεδρε, να κρατήσετε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίρρηση ότι θα αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Η κυρία Σίνοτ. Υπάρχει λόγος που η Κομισιόν θα πρέπει να διερευνήσει το θέμα αυτό πολύ σοβαρά. Ο συνάδελφός μου σας εξήγησε γιατί. Τι συνέβη σε αυτήν την περίπτωση. εργολάβοι ή τα αεροδρόμια ή αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τις κοινοτικέ ε, οδηγίες για να παλωτριώσουν γη και για να παλωτριώσουν τους ιδιοκτήτες από τα ιδιοκτησιακά τους ε, δικαιώματα. Ίσως ε, δεν θα είχαν γλιτώσει αν είχε ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί ο κόσμος θα ήθελε να έχει ενημερωθεί. Θα ήθελε να δει επιστημονικά στοιχεία για αυτές τις ζώνες ασφαλείας. Αλλά και δεν θα είχαν ευκαιρία λοιπόν να τους αρπάξουν τη γη. Από την άλλη υπάρχουν και παραδείγματα άλλων περιπτώσεων αναφορών που φτάνουν στην Επιτροπή Αναφορών, όπου ε, ουσιαστικά κροϊδεύουν την κοινωνία των πολιτών. Θέλουν να αρπάξουν τη γη, α πούμε, και κρατάνε μυστικά. Υπάρχει ένα πολύ επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τι κοινωτικέ οδηγίε. Αν θέλουν κάτι και του βολεύει, τι λένε αμέσω, Α, η Ευρώπη το θέλει χρησιμοποιούν αυτό που θέλουν, παίρνουν αυτό που θέλουν. Κάνουν ό,τι μπορούν για να αρπάξουν αυτό που θέλουν. Και νομίζω ότι αν η Κομισιόν δεν διερευνήσει πολύ σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικέ αρχέ, η Ιρλανδική κυβέρνηση και όλοι οι λοιποί που πούμε, ασχολούνται με την ιδιοκτησία του κόσμου, με τους κινδύνους που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές, νομίζω ότι θα έχουμε όλο και περισσότερο απογοητευμένους εκλογής. Προέδρο. θα σου Πρόεδρος, άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Η Κομισιόν έχει να πει τίποτα. Μια και οι επικρίσεις αφορούν και την Επιτροπή τελικά. Οι Ιρλανδοί βουλευτές θεωρούν ότι υπάρχει παράβαση. Μήπως η Κομισιόν θα ήθελε να σχολιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία σε Βέζο έχει ως σκοπό να προστατεύσει τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υποστούν ατυχήματα, μεγάλα ατυχήματα. Και επομένως ε, υπήρχαν και αυτές οι διατάξεις για το σχεδιασμό ε, ανάπτυξης κάποιων χώρων. Τώρα, η εφαρμογή γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα για αξιολόγηση του κινδύνου και αυτό είναι θέμα που το καλύπτει η εθνική νομοθεσία. Δεν είναι θέμα της Ευρώπης. Αυτός ο σχεδιασμός και οι σχετικές διατάξεις απαιτούν ε, μία αξιολόγηση του κινδύνου για τις νέες εγκαταστάσεις. Και η πιο σημαντική διάταξη αυτής της οδηγίας είναι αυτό το άρθρο που μιλάει για αυτό το σχεδιασμό. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Κάναμε μια προσπάθεια να εναρμονίσουμε την αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη και να εφαρμοστεί σωστά το σχετικό άρθρο. Όπως σας εξήγησα, όμως η οδηγία αυτή καθεαυτή μιλάει για την υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους μεγάλους κινδύνους και ατυχήματα όταν σχεδιάζουν ε, το πώς θα χρησιμοποιήσουν ε, τη γη και τι εγκαταστάσει θα κατασκευάσουν κτλ οι εφαρμοστικές ευθύνες ε, βαραίνουν τα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται όλα αυτά πώς τα κράτη-μέλη. Είναι θέμα κρατών μελών. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αναφέροντα σε αυτό το σημείο, γιατί η οδηγία αφορά τις νέες εγκαταστάσεις μόνο. Δεν μιλάει για Ολε τι εγκαταστάσει και όλα τα θέματα σχεδιασμού στα κράτη-μέλη, σχεδιασμού αυτών των εγκαταστάσεων. Πρόεδρο. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ πλήρω. Άλλο είναι να πούμε ότι ο αστικό σχεδιασμό είναι θέμα ευθύνη του κράτου μέλου και τελείω διαφορετικό το να πούμε ότι οι συνέπειε αυτού του σχεδιασμού παραβιάζουν τις, ε, την κοινοτική νομοθεσία και τι κοινοτικέ αρχέ. Αυτό το δεύτερο είναι δική μα αρμοδιότητα η παραβίαση. Αν λέγαμε, ας πούμε, ότι ο αστικός σχεδιασμός ήταν αποκλειστικής αρμοδιότητας του, των κρατών μελών, τότε δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ασχοληθεί με τα ισπανικά θέματα, ούτε θα είχαμε συζητήσει την έκθεση Άουκεν, την οποία ψηφίσαμε και υιοθετήσαμε πριν από λίγο. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μου πει αν έγινε αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου. Και αν ξέρετε τα αποτελέσματα αυτής της ε, έρευνας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία υιοθετήθηκε το 1996. Τότε δεν είχαν γίνει, ούτε απαιτούνταν να γίνουν αξιολογήσεις του κινδύνου. Και δεν υπήρχαν σχετικά έγγραφα, λοιπόν. πρόεδρος. Επομένως, θα πρέπει να γράψουμε μια πολύ αυστηρή επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο της Ιρλανδίας και να εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η άποψή μας. Και να ζητήσουμε να μας εξηγήσει το Υπουργείο την άποψή του και τη στάση του. Δεν είναι μια λύση προς το πρόβλημα, είναι ένα βήμα στην όλη διαδικασία. Θα, θα ήθελα να μου πούν οι αναφέροντες αν τους ικανοποιεί αυτή η λύση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λυπάμαι που η Κομισιόν νύπτει τα σχήρα τη, γιατί η οδηγία αφορά και τις ισχύουσες εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία. Τέλος, ο τρόπος που εφαρμόστηκε στα αεροδρόμια και στις περιοχές σε Βέζο δεν ήταν σωστός. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα ασφάλειας. Και επομένως ε, Υποστηρίζω την αναφορά Γκίλιγκαν. Ε, υποστηρίζω τα όσα είπατε. Προσοχή, Πρόεδρε, γιατί ε, ο κόσμος θα αποθαρρυνθεί και θα αποστραφεί από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Γαλλία έγινε σωστά. Ε, εφαρμόστηκε σωστά αυτή η οδηγία. Θέλουμε να δούμε τι έγινε στη Γαλλία. Θα πρέπει ε, οι εταιρείε όπως η ΡΑΣ να αποζημιώσουν τον κόσμο στην Ιρλανδία υπάρχει ε, σωστή χαρτογράφηση των ζωνών σε βέζο. Δεν γνωρίζουμε ποιε είναι αυτέ οι καταστάσει σε βέζο. Το λέμε στο κείμενο. Να, ποια είναι η γη του κ. Γκίλιγκαν, με πράσινο. Ε, υπάρχουν πέντε ζώνες ασφαλείας πάνω στη γη του και ποτέ δεν ενημερώθηκε ε, για την ευκαιρία που θα έχει να κάνει κάποια διαβήματα. Δύο από αυτέ τι ζώνες είναι σε Βέζο και τρει είναι ζώνε ασφαλεία αεροδρομίου. Ποτέ δεν είχε την ευκαιρία να κάνει καμία προσπάθεια, κάνει ένα διάβημα α πούμε καμία αναφορά σε εφημερίδα ότι θα επιβληθεί μια ζώνη σε Βέζο. Μας είπαν απλώς ότι το, ε, οι δημοτικές αρχές θα αλλάξει ας πούμε, τον τρόπο σχεδιασμού. Δεν υπήρχε καμία διαφάνεια. Αυτά, Πρόεδρε, σας παρακαλώ να διερευνήσετε το θέμα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό που είπα. Θα γράψω μια επιστολή στο Υπουργείο και θα ζητήσουμε μια εξήγηση. Θα ήθελα να μας σχολιάσει λοιπόν το Υπουργείο ε, όλα αυτά που αναφέραμε και τι έχει να πει για τις κατηγορίες μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή. Proszę Państwa, ponieważ myśmy zapowiedzieli, że raport pani e, Diany Wallis... Επειδή λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Βόλης ε, την έχουμε προβλέψει ε, για τις 12 και 12, να μην τα μπερδέψουμε, μην δημιουργήσουμε χάος και γι' αυτό προτείνω να ασχοληθούμε τώρα με το 28 μετά με το 29 και γύρω στις 12 ε, και 4 να πάμε πίσω στην ε, τοποθέτηση της κυρίας Γουόλτ. Λοιπόν, 28, ε, αναφορά του 2006, η Κομισιόν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα μέσα σε δύο λεπτά να σας παρουσιάσω μια γενική προσέγγιση όσον ε, αφορά στην προσπάθεια της Κομισιόν να επιβάλλει κάποια ποιότητα με βάση οδηγίες. Γιατί στην ημερήσια διάταξη έχουμε τουλάχιστον τέσσερις συναφείς ε, αναφορές. Όσον αφορά λοιπόν σε αυτή τη γενική προσέγγιση, θέλω να πω το εξής. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ε, ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξαν υπερβάσεις. Η Κομισιόν λοιπόν εκλήθη επανειλημμένα να μας πει τι θα κάνει Λοιπόν, η Κομισιόν κατέληξε στο ότι αντί να επιβάλλει σε 26 κράτη-μέλη μία άποψη, θα πρέπει να βρεθεί ένα νομικό εργαλείο για να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα. Και μέχρι το 2008 ε, μάλλον το 2008 τέθη μια νέα οδηγία σε ισχύ και αυτή η οδηγία εξετάζει ακριβώς αυτές τις ε, υπερβάσεις ε, επικυρώνοντας τα όρια, προσφέροντας όμως και τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν, να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις ε, της οδηγίας. Η Κομισιόν κατόπιν έστειλε μια επιστολή πριν από την επίσημη όπου ενημέρωσε τα κράτη-μέλη για την υποχρέωσή τους να ε, συμφωνήσουν, να συμβαστούν με τις οριακές τιμές και είτε να ζητήσουν παράταση χρόνου ή εν πάση τόση να ε, συμβαστούν όπως ε, είπαμε με τις οριακές τιμές και αυτά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2008. Πήραμε λοιπόν κοινοποίηση από 13 κράτη-μέλη και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση αξιολόγησης των ετοιμάτων τους. Αλλά από 10 κράτη-μέλη δεν πήραμε καμία κοινοποίηση ε, σε σχέση με, το, με την με το συμβασμό τους με το PM10 ή εν πάση περιπτώσει δεν μας ενημέρωσαν για τους τομείς στους οποίους υπάρχει υπέρβαση. Ε, κατά τα τέλη λοιπόν Ιανουαρίου αρχίσαμε τη διαδικασία επιπαραβάση εις βάρος 10 κρατών μελών. Ως εκ τούτου, επειδή σας τα είπα έτσι κάπως γενικότερα, θα ήθελα τώρα να επανέλθω στις συγκεκριμένες αναφορές. Λοιπόν, πάμε στην 959. Σε μία, με μία μονοπρόταση θα μπορούσα να πω το εξής. Εδώ ε, πρόκειται για την ε, μόλυνση του περιβάλλοντος και την, ε, τον θόρυβο στην Μάλτα λόγω του εργοστασίου το οποίο αποκαλείται Blockrit LTD. Εδώ ισχύουν κάποιοι κανόνες και αφορούν βεβαίως και τη λειτουργία αυτού του εργοστασίου ζητήσαμε από την αρμόδια αρχή να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Δηλαδή το πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση, ε, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η δυσαρέσκεια. Είπανε ότι η εθνική επιθεώρηση προβαίνει σε κάποιες ενέργειες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εδόθησαν λεπτομέρειες για τα μέτρα που λήφθησαν. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήθελα να πω ότι η οδηγία περί θορύβου, αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θόρυβο, δεν ισχύει καθότι περιορίζεται μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα και όχι σε μικρές πόλεις ή μικρές εγκαταστάσεις. Πάντως, όσον αφορά την ενόχληση σχετικά με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, γνωρίζουμε ότι η πόλη αυτή βρίσκεται σε μία περιοχή η οποία επίσημα ανακηρύχθηκε ως περιοχή που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια αιωρούμενων σωματιδίων. PM10 όπως αποκαλούνται. Η Κομισιόν λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, αξιολογεί το πρόγραμμα ποιότητας που έχει εκπονήσει. Και στην ε, προηγούμενη φάση, την προαξιολόγηση, σε, ε, αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένα μέτρα για το εργοστάσιο blockreed Εντοπίσαμε και κάποιες άλλες αδυναμίες. Επανήλθαμε λοιπόν στα κράτη-μέλη έτσι ώστε ε, να βοηθήσουν να υπάρξει μια τεχνική αξιολόγηση και να ληφθεί μια απόφαση όπως ακριβώς προβλέπεται από το άρθρο 22. Ε, η Μάλτα βέβαια είχε ενημερώσει έγκαιρα και ως εκ τούτου αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνεται στα 10 κράτη-μέλη τα οποία έχουν οδηγηθεί στην διαδικασία επιπαραβάση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλήσαμε τελευταία φορά για αυτή την αναφορά ήταν το 2007. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα πράγματα όσον αφορά τις συγκεκριμένε εξελίξεις στο θέμα αυτό από αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να πω ότι η κατάσταση αυτή, σε αυτή την ειδική κατάσταση όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά, ε, έχει αποδειχθεί. Εγώ ίδια επισκέφθηκα αυτή την επιχείρηση, υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, αλλά δεν επαρκούν και είναι συνεπώς βάσιμη αυτή η αναφορά. Και θα πρέπει να πω ότι έγιναν πολύ περισσότερες καταγγελίες που έφτασαν στα χέρια μου και ξέρω ότι έχουν υποβληθεί και άλλες αναφορές όσον αφορά και άλλες περιοχές από τη Λύχια, την Ασάρ, το Σιτζίουι. Πολλές από αυτές τις ε, αναφορές θα φτάσουν τελικά στα χέρια μας. Την τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, που συναντηθήκαμε σχέση με αυτή την αναφορά, είχα ζητήσει ειδικά από την Επιτροπή, από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, να μας ε, παραπέμψει ένα κατάλογο ε, ε, υποχρεωτικών μέτρων τα οποία θα έπρεπε να επιβάλλουν οι εθνικές αρχές σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Και επίσης να επανέλθει σε εμά υποβάλλοντας ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το πότε θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα υποχρεωτικά μέτρα. Και πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μας δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο να κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πραγματικά θα έπρεπε να έχουμε τώρα μια απάντηση και θα ήθελα να κλείσω εδώ γιατί νομίζω ότι η Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να μας δώσει μια απάντηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Ναι, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Και Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω το εξή. Πράγματι, δεν γνωρίζω εάν η Κομισιόν επιθυμεί να σχολιάσει, αλλά εάν ε, υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρου του κυρίου Μπούσουτιλ ε, που διατυπώθησαν παρουσία του εκπροσώπου της Επιτροπής, είναι κρίμα που η Επιτροπή δεν απάντησε. Θα πρότεινα να σχολιάσει γραπτά η Επιτροπή το θέμα αυτό εντός δύο εβδομάδων. 29. Πρόκειται για την αναφορά 1232 του 2007. Ο κύριος Μανουέλ Γαρθία Γκονζάλες είναι ε, παρόν και επίσης και ο αρμόδιος υπουργός Εξερμαδούρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω θερμά τον αναφέροντα καθώς και τον κύριο υπουργό και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Ε, buenos días. 5 minutes. Έχετε πέντε λεπτά. Ε, Καλημέρα σας. Ε, θα εκπροσωπώ τον κύριο Μανουέλ ε, Ροδρίδε, ο οποίο δεν μπόρεσε να παραστεί. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μας δώσετε τη δυνατότητα να παρέμβουμε σε αυτό το φόρουμ. Συγγνώμη, θα επαναλάβω. Πέτρο Βισέντε Σάντσοφ εκ μέρους της πλατφόρμας των πολιτών. Πλατφόρμα Σεροδάνα Ρεφενερία. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ που μας δώσετε τη δυνατότητα να παρεύουμε σε αυτό το σώμα εκπροσωπώντας ένα ιδιαίτερο σημαντικό τμήμα της κοινωνίας της Ανταλουσίας που είναι αντίθετο προς το πρόγραμμα εγκατάστασης ενός δηληστηρίου που θέλουν να επιβάλλουν οι ισπανικέ αρχέ στου πολίτε τη Ισπανία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο πρόθεσε ο κύριο Αλφόνσο Σογκαλιάρδο, ένα επιχειρηματίας ο οποίο έχει κατηγορηθεί πολλέ φορέ ότι επιβαρύνει με εξαγλωριούχο βενζένιο ε, την ατμόσφαιρα τη Ισπανία και είναι ο μεγαλύτερο ρηπαντή σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά αυτή την τοξική ουσία. Ε, το Πρόκειται για την εγκατάσταση ενός διαχειριστηρίου ε, πετρελαίου ε, σε μια χώρα όπου έχει 3.000 ε, χιλιόμετρα ακτογραμμή. Το αργό πετρέλαιο πρέπει να μεταφερθεί μέχρι το λιμένα της Ουέλβα και θα πρέπει να διανύσει συνεπώς 250 χιλιόμετρα έως ότου φτάσει σε ένα ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πάνω από 400 μέτρα. Και με τον τρόπο αυτό θα δαπανηθεί το 7% του συνόλου της ενεργειακής δαπάνης της, του εργοστασίου. Πέρα από αυτό... Ε, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η πρόθεση να εξαχθούν τα προϊόντα του διελισμού, ενώ η, τεκμηρίωση αυτού του προγράμματος ε, λέει ότι είναι, οφείλεται στην έλλειψη, ανάγκη στην έλλειψη πετρελαίου στην Ισπανία. Όλα αυτά οδηγούν σε μια αυξημένη κίνηση πετρελαιοφόρων και φορτικών ε, πλοίων που είναι περίπου 200 κάθε χρόνο ε, και προστίθενται στα φορτηγά τα οποία κυκλοφορούν κοντά στην ακτή της ε, Ουέλβα και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι επιβαρύνονται 11 οικότοποι της περιοχής, δηλαδή το Πάρκε Νασιονάλ Ντονιάννα. Ε, το διελιστήριο αυτό πρόκειται να εγκατασταθεί σε μία από τις πιο αφορές περιοχές της Εξτρεμαδούρα που λέγεται Τιέρα Ντεμπάρος και όπου απασχολούνται 20.000 ε, εργαζόμενοι. Από την άλλη ε, θα πρέπει να αντλούν τεράστιες ποσότητες υδάτων το χρόνο σε μια ζώνη που χαρακτηρίζεται τα λειψιδρία από χαμηλές βροχοπτώσεις και τα ύδατα αυτά θα πρέπει να αντλούνται από τα αποθέματα του ποταμού Γουαδιάνα με τον τρόπο αυτό απειλώντας τα αποθέματα του ποταμού και ρηπαίνοντας ε, τα νερά του με τον τρόπο αυτό ζημιώνοντας και τα συμφέροντα της Πορτογαλίας γιατί στην επικράτεια της Πορτογαλίας εκβάλλει τελικά ο ποταμός αυτός ο Γουαδιάνα. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορα οικονομικά προγράμματα της Πορτογαλίας για την ανάπτυξη της περιοχή τη Αλκουέβα. Το πρόγραμμα αυτό ε, στοχεύει στην συγκράτηση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του Αλάγκε και αυτό θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον γιατί η περιοχή αυτή είναι τμήμα της ζώνης ειδικής προστασίας για τα πτηνά. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζει η Οδηγία 79409 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου σε σχέση με την προστασία των πτηνών. Ε, τα σχέδια τα οποία προβλέπονται για το πρόγραμμα αυτό και άλλα σχέδια κατασκευής κεντρικών θερμοελεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η των νερών από το ποταμό Γουαδιάνα ε, αντιβαίνουν στο πνεύμα της ε, Οδηγίας 2060 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23 Οκτωβρίου του 2000 ε, δια της οποίας θεσπίζεται το κοινοτικό πλαίσιο προστασίας των υδάτων και στην οποία αναφέρονται το άρθρο 1, 5 και 9 και ειδικά το άρθρο 12 σε σχέση με τα προβλήματα που φορούν όχι μόνο μια χώρα μέλος αλλά περισσότερες χώρες δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του ποταμού Γουαδιάνα. Ε, επιπλέον δεν έχει γίνει καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όλα αυτά αντιβαίνουν στην οδηγία που σας ανέφερα και που αφορά την ενημέρωση του Συμβουλίου. Γιατί δεν δόθηκαν επίσης, δεν δέθηκαν στη διάθεση των Ισπανών πολιτών τα στοιχεία σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Μόνο εκ των υστέρων παρουσιάστηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το δηληστήριο αυτό και το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε με τρόπο ε, Δεν ε, δόθησαν αντίγραφα στους πολίτες που το ζήτησαν. Με τον τρόπο αυτό σημειώθηκε μια παραβίαση ε, του χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η πλατφόρμα των πολιτών, την οποία εκπροσωπούμε, δεν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους δημόσιους χώρους για τις συναντήσεις της. Παρακαλώ να καταλήξετε γιατί ε, θα πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, η εκπρόσωπο της Επιτροπής παρακαλώ να είναι σύντομη στην παρουσίασή της. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή προσεκλήθη στην Επιτροπή αυτή για να παρουσιάσει τη δική της άποψη σε σχέση με την υπόθεση αυτή που με την οποία ασχολήθηκε η Κομισιόν λόγω γραπτών αναφορών όπως αυτή την οποία συζητούμε σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρχές ε, σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα και ε, τονίσαμε την ανάγκη να τηρούνται οι σχετικές οδηγίες για το περιβάλλον. Υπό την έννοια αυτή και σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, το εν λόγω πρόγραμμα ε, έχει υποβληθεί σε μια διαδικασία εξολόγηση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σύμφωνα με την ε, οδηγία που καλύπτει τη διαδικασία αυτή. Και Φόσον γίνει η εξολόγηση του προγράμματος αυτού, θα υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών και διαβούλευσης. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να πούμε ότι η οδηγία με τα άρθρα 6 και 7 αναφέρει την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού και έναρξης κάποιων ε, διαδικασιών ε, διαβούλευσης με το κοινό που θα πρέπει να τηρούνται από τις χώρες μέλη και ή δυνατόν θα πρέπει να τηρούνται αυτές οι γενικές αρχές. Πρόκειται για κάποιες αρχές που λαμβάνει υπόψη της Επιτροπή για να μπορέσει να διαπιστώσει εάν γίνονται σεβαστές οι διατάξεις της οδηγίας. Οι πολίτες σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και θα πρέπει να έχουν επίσης την δυνατότητα σε εύλογο χρόνο να μπορέσουν να παρουσιάσουν γραπτά σχόλια θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τηρούνται τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες και ενημέρωση των πολιτών. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη αυτών των, για τον τρόπο που έγιναν αποδεκτά αυτά τα γραπτά σχόλια. Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται και να έχουν πρόσβαση επίσης στα ένδικα μέσα προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ε, ε, σύμφωνα με την αναφορά αυτά, αυτή ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις, αλλά ε, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια προσφυγή στα ένδικα μέσα της Ισπανίας στην ελόγω περίπτωση. Το πιο σημαντικό για την περίπτωση αυτή είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό για το δηληστήριο. Η Κομισιόν δεν έχει στη διάθεσή της επαρκή δεδομένα για να σας πει κατά πόσο πρόκειται εδώ για μια παραβίαση, κατάφερε παραβίαση του κοινωτικού δικαίου. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός της Εστρεμαδούρα θα πάρει το λόγο και εν συνεχεία οι βουλευτέ. Και μετά κλείνει ο κατάλογος των υπουργών. Ο υπουργό, ο κ. Σέρκα, ο κ. Μέγερ και ο κ. Χάμερστάιν Μίντς. 1,5 λεπτό καθένα, παρακαλώ. Buenos días. Καλημέρα σα, σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε δυνατότητα να παρέμβω εκπροσωπώντας την ε, Περιφερειακή Κυβέρνηση Εξτρεμαδούρα για να σας εξηγήσω πώ θεωρούμε ότι η διαδικασία αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος εγκατάσταση δηληστηρίου εξελίσσεται ε, τηρώντας αυστηρότατα τι διατάξει οδηγίες όσον αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώ και τη δυνατότητα πρόσβαση εκ μέρου των πολιτών σε πληροφορίε. Το πρόγραμμα του δηληστηρίου αξιολογείται εκ μέρους της ε, κυβέρνησης της Ισπανίας. Το αρμόδιο όργανο είναι το Υπουργείο της Βιομηχανίας και το όργανο που αφορά το περιβάλλον είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ε, έχουν υποβληθεί τα στοιχεία αυτά στο κοινό και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πρόγραμμα στην Ισπανία, δημόσιο ή ιδιωτικό, το οποίο να συνδέεται πρώτα σε εγγύηση συμμετοχή εκ μέρου των πολιτών. Η μεταφορά τη οδηγία στο Ισπανικό Δίκαιο προποθέτει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται αυτή η πρόσβαση στις σχετικές ε, πληροφορίες και ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω ίντερνετ. Ε, και μάλιστα οι ισπανικέ Αρχές έθεσαν ε, στη διάθεση των πολιτών μία αίθουσα με υπολογιστές, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες για να αντλήσουν αυτά τα στοιχεία. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των αρχών, οι αμφιβολίες αυτές ε, λύθηκαν υπό την έννοια της παροχής περισσότερων εγγύσεων. Γιατί ξέραμε ότι η δεξία αυτή πρόκειται να υποβληθεί σε έναν πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο. Όσον αφορά την ε, διασυνοριακή εφαρμογή, στην τελευταία ε, συνάντηση κορυφής μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, ε, ο Πορτογάλος Υπουργός Περιβάλλοντος έθεσε, παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό σαν ένα υποδειγματικό πρόγραμμα καλή συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών μελών όσον αφορά θέματα διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όσον αφορά το θέμα των υδάτων, η άντληση νερών ε, αφορά τη λεκάνη απορροής του ποταμού αυτού του Γκουαδιάνα και που ενδιαφέρει τόσο την Ισπανία όσο και την Πορτογαλία. Θα ήθελα να πω ότι η ποσότητα των υδάτων που αντλούνται αντλούνται από μια περιοχή όπου τα ύδατα είναι επαρκή τόσο για τις γεωργικές ε, καλλιέργειες όσο και για την, ε, το, την άντληση του πόσιμου νερού. Ε, όλες οι καταγγελίες υποβλήθησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο τις μελετά και θα απαντήσει. Εξάλλου πρόκειται να διενεργηθεί μια έρευνα ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και τώρα θα ήθελα να σα πω κάποια άλλα στοιχεία για την εξερμαδούρα. Πρόκειται για μια περιοχή όπου έχουμε μόνο 26 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο όπου υπάρχει ανεργία της τάξης του 18%, όπου ο βιομηχανικός τομέας είναι 6% σε σχέση με το 13% του συνόλου της Ισπανίας και ένα ΑΕΠ σε σχέση με το ευρωπαϊκό των 27% του, που είναι 70% του συνόλου της Ευρώπης. κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών ε, αυξήθηκαν σημαντικά οι θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να σας πω ότι η θέση της περιφερειακής κυβέρνησης είναι να δείξει πλήρη εμπιστοσύνη προ όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε σχέση με την απόφαση που θα ληφθεί τελικά, όποια και είναι αυτή. Γιατί κατανοούμε ότι τα πράγματα γίνονται μεν ε, καλώ, αλλά θα ήθελα να πω ότι για την περιοχή τη Εξτρεμαδούρα, εάν ε, στην Ισπανία εγκαθίσανε διάφορα διελιστήρια πετρελαίου με περιβαλλοντικές επιπτώσεις ισότιμες με αυτήν αυτής της περιοχής, δεν κατανοούμε γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Εξερμαδούρα ενώ επιτρέπεται σε άλλες περιοχές της Ισπανίας. Ο κύριος ε, Παντσέρκας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, Ακούσαμε τις γνώμες της πλατφόρμα, τις γνώμες του Υπουργού, τις γνώμες άλλων συναδέλφων. Η δική μου περίπτωση είναι η διάζουσα. Εγώ είμαι ένας βουλευτής αυτής της περιοχής, εκεί πέρασα την παιδική μου ηλικία, την νεότητά μου και γνωρίζω απολύτως τα στοιχεία. Και θα ήθελα απλώς προκειμένου να αξιολογηθεί το θέμα αυτό με προσοχή και ακρίβεια, γιατί εδώ πρόκειται για μια πολιτική συζήτηση, θα πρέπει να γνωρίσουμε δύο θεμελιώδη θέματα. Όσον αφορά το επιχείρημα ότι ε, θα πρέπει να γνωρίσω ότι όλοι οι πολιτικοί είναι υπέρ, που εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο, στο περιφερειακό κοινοβούλιο της περιοχής, είναι υπέρ της εγκατάστασης του δηληστηρίου στην Ισπανία έγιναν ε, εκλογές ε, στα χωριά αυτά ε, και ρωτήθηκαν οι κάτοικοι και παντού η απάντηση ήταν καταφατική υπέρ του διαλυστηρίου. Η κοινή γνώμη στη δική μου περιοχή που είναι μια περιοχή η οποία χρειάζεται απασχόληση, είναι πολύ στατική υπέρ της εγκατάστασης του διαλυστηρίου και αυτοί είναι οι πρωτίστως ενδιαφερόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτή η μελέτη. Συνεπώς, κανείς δεν εξουσιοδοτείται να μιλήσει εξ ονόματος της φύσης, εφόσον η έρευνα αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους αναφέροντας και θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και με τις πληροφορίες που κόμισαν εδώ οι αναφέροντες, η αναφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή ε, λόγω της βαρύτητας αυτού του έργου ε, και λόγω του μεγέθους της ε, ακτογραμμής στην περιοχή αυτή. Εδώ πρόκειται και ένα θεμελιώδες θέμα. Νομίζω θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια σφάλματα που αφορούν τη συμμετοχή των πολιτών. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ της Πορτογαλικής και Ισπανικής αρχής, γιατί στην Πορτογαλία είχαν η δυνατότητα οι πολιτικές ομάδες και οι κοινωνικές ε, ενώσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, ενώ αυτό δεν έγινε στην Ισπανία. Οι πολίτες θεωρώ ότι δικαιούνται να έχουν τα πλήρη, τις τα πλήρη στοιχεία σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό και θεωρώ κύριε Πρόεδρε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση του προγράμματος πολύ σημαντική και θα πρέπει αναφορά αυτά να παραμείνει ανοιχτή ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει συνεχεία και αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Το να εγκατασταθεί μια, ένα δηληστήριο σε μια τέτοια περιοχή στην ενδοχώρα ε, είναι παράλογο γιατί όλα τα δηληστήρια βρίσκονται σε παράκτες περιοχές για προφανείς λόγου. Είναι σαν, ε, λόγους. Είναι σαν να φτιάχνουμε ένα χιονοδρομικό κέντρο εν μέσω της Σαχάρας θα πρέπει η Επιτροπή να μην περιορίζεται να επαναλαμβάνει ποιοι είναι οι νόμοι, οι διατάξεις και να μην απαντάει ποτέ. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν ε, μελετάει τις σορευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όχι μόνο του ιδίου του δηληστηρίου, γιατί στην ίδια ζώνη υπάρχουν ε, θερμοελεκτρικές εγκαταστάσεις, υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής ε, τσιμέντου και νομίζω ότι θα πρέπει να μελεθούν συνολικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά δεύτερο λόγο, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, δεν θα πρέπει να εξετάζει, να περιορίζεται μόνο στην πόλη της ε, Ουέλβα, χρησιμοποιώντας συγκριτικά στοιχεία που αφορούν μόνο την πόλη αυτή, η οποία είναι από τις πιο μολυσμένες πόλεις του πλανήτη. Ε, τα πετρελαιοφόρα θα πρέπει να διανύουν ε, από τις πιο όμορφες περιοχές της Ισπανίας, βορείως της ε, Ουέλβα, από εκεί που προέρχεται για παράδειγμα το περίφημο ζαμπόν του Μπανδούγο. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρος, είναι προφανές ότι παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά τη στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει ότι δεν έχει ε, καθοριστικά και ε, τελεσίδικα στοιχεία. Θα επιληφθούμε λοιπόν του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε τον αναφέροντα και τον κύριο Υπουργό από την Εστρεμαντούρα και επανερχόμεθα στη γνωμοδότηση, στην τοποθέτηση της κυρίας Γόλης σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν. Κυρία Γόλης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και επίσης ε, σας ευχαριστώ πολύ που ε, μου δίνετε το χρόνο για να παρουσιάσω την έκθεσή μου. Είναι μια έκθεση που κάνουμε κάθε χρόνο. Μετά από την ε, έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση του κοινοτικού δικαίου. Τη βασική έκθεση την κάνει η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Συνεργαστήκαμε με τον ε, εισηγητή σε αυτήν την Επιτροπή. Είναι η δεύτερη τρίτη φορά που κάνω αυτή την έκθεση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γράφω κάποια από τα σχόλια που διαβάζετε στην εκθεσή μου. Είναι θλιβερό αυτό. Γιατί θα ήθελα να αισθάνομαι ότι γίνεται πρόοδος. Συχνά σε αυτή την Επιτροπή βρισκόμαστε στις, στους προμαχώνες όπου παρακολουθούμε πώς λειτουργεί το κοινωτικό δίκαιο και τι προσφέρει στους πολίτες. Κάποια πράγματα λοιπόν που διαβάζετε τα έχω ξαναπεί πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη οι πολίτες μας να πλησιάζουν τα θεσμικά όργανα με απλό τρόπο όταν πιστεύουν ότι κάτι είναι σφαλμένο ή δεν λειτουργεί. Πιστεύω ότι ε, είχαμε πάντα εκφράσει την ε, ιδέα ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία μόνο απευθυντική θηρίδα, ούτως ώστε να απευθύνονται σε αυτή την ε, θηρίδα η Επιτροπή, στον Επιτροπή μας, στον Διαμεσολαβητή ή στο Solvit. Τώρα πάνε μάλλον στο Διαμεσολαβητή, στο Solvit κτλ. Η κατάσταση είναι... προκαλεί συγχύσεις. Θα πρέπει να τη διευκολύνουμε την κατάσταση για τους ε, πολίτες. Ούτως ώστε η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου να είναι πιο αποτελεσματική Πώς θα το κάνουν τα φέρουν αυτό οι πολίτες αν δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Επομένως αυτή η θηρίδα παραμένει μία από τις προτεραιότητές μας. Επίσης, θα ήθελα να μας πει περισσότερα πράγματα η Επιτροπή για το πώς ε, ερμηνεύει την ευθύνη του ευθύνη, ε, ερμηνεύει μάλλον την ιδέα του, της κρατικής ευθύνης σε, σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Θα ήθελα κάτι πιο απτό για αυτό το θέμα μπροστά μας. Τώρα θα ήθελα να σχολιάσω δύο τομείς που αλληλοσυνδέονται και που ενοχλούν πάρα πολύ αυτή την Επιτροπή. Εμείς είμαστε βουλευτές, αλλά παράλληλα είμαστε και πολίτες. Και όταν υπάρχει διάλογος μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών για μια πιθανή παραβίαση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού του διαλόγου. Τώρα είναι τα πράγματα απόλυτα συγκεχημένα ως το τι συμβαίνει ανάμεσα στην Κομισιόν και στο, στα κράτη-μέλη. Και σε εμά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και το πρόβλημα είναι ότι συχνά η απόφαση είναι πολιτικού χαρακτήρα για το αν θα ξεκινήσει μία διαδικασία επί παραβάση. Ίσως είναι τμήμα ε, ενός πακέτου, ε, μια συμφωνίας που κάνουν τα κρατη με την Κομισιόν. Αλλά αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για μας, ούτε για τους πολίτες. Για αυτούς που είναι οι αποδέκτες της νομοθετικής δουλειάς. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό όταν υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και έχει γίνει ζημιά επίσης. Και ο πολίτης ή οποιοδήποτε είναι αυτός γνωρίζει ότι έχει υπάρξει παραβίαση και η Κομισιόν καταλήγει δικαίως ή αδίκως στο συμπέρασμα ότι έχει σταματήσει η παραβίαση αλλά το άτομο αυτό ή ο φορέας κτλ. Ε, έχει υποστεί τη βλάβη ούτως ή άλλως και συχνά δεν υπάρχει αποζημίωση ή διόρθωση του προβλήματος. Ή συχνά, αν υπάρχει αποζημίωση, ε, η διαδικασία είναι πάρα πολύ περίπλοκη, πάρα πολύ δεδαλώδης και δαπανηρή, όπως ε, είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως μία που ξέρω πολύ καλά που αφορά την υπόθεση του Equitable Life. συχνά αναφέρουν κάτι οι πολίτες, υπάρχει παραβίαση, γίνεται κάτι για να σταματήσει η παραβίαση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αποζημίωση, υπάρχει ε, επανόρθωση της βλάβης. είναι το πρόβλημα. Γίνονται πολλά πράγματα για να βελτιωθεί το σύστημα, για να γίνει πιο διαφανές, το αναγνωρίζουμε αυτό και είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό, ότι δηλαδή στην ε, αρχή της ζωής ενός νομοθετήματος, ε, συχνά ε, υλοποιούνται τα αιτήματα των πολιτών μέσα από τα λεγό, τις λεγόμενες συνόψεις των πολιτών. Ε, μα αυτές τις συνόψεις καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και αν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται καταλαβαίνουμε και τι δεν πάει καλά. Καλό είναι λοιπόν που προοδεύουμε σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να κάνουμε πολλές ακόμα προσπάθειες και αυτές οι συνόψεις, οι περιλήψεις των πολιτών παραμένουν στο επίκεντρο της διαδικασίας και όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Στην έκθεσή μας επίσης λέμε κάτι και εδώ συμφωνούμε με την Κομισιόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Να υπάρχουν πίνακες επαλήθευσης όταν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την ε, κοινοτική νομοθεσία, τη μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δούμε πώς ακριβώς την εφάρμοσε, τι ακριβώς έχει συμβεί. Συχνά το Κοινοβούλιο είναι ένοχο ε, ως συνομοθέτης επειδή δεν ήταν αρκετά αυστηρό. Επειδή δεν παραμένουν στα νομοθετικά κείμενα αυτοί οι πίνακες επαλήθευσης. Εγώ με ανησυχία παρατήρησα πολλές συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης στο πρόσφατο παρελθόν και στην πραγματικότητα τι συνέβαινε, ότι εμείς αυτές τις συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης είχαμε παραιτηθεί από αυτούς τους πίνακες επαλήθευσης. Η Κομισιόν όμως πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Πάντα τους προτείνει αλλά εμείς δεν επιμένουμε ή και το Συμβούλιο δεν επιμένουμε μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Θα πρέπει να το κάνουμε αν είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Τώρα κάποια γενικά σχόλια. Μέσα σε αυτή την απογοήτευσή μας, το ακούσαμε και σήμερα το πρωί, μέσα στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι θα πρέπει οι πολίτες συλλογικά να έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια με έναν οικονομικό και εύκολο τρόπο. Έχουμε προτάσεις στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού και στον τομέα του δικαίου περί καταναλωτών αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. κάτι, κάποια κράτη-μέλη, ένα από αυτά είναι η Πορτογαλία, που λείτες πολύ περισσότερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση συλλογικά, σε συλλογικές προσφυγές στα δικαστήρια. Όταν μια ομάδα ανθρώπων έχουν υποστεί ζημία. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι σε πολλούς τομείς. και μπορεί να γλιτώσουμε και ένα μεγάλο αριθμό αναφορών, αν και πάντα χαιρόμαστε να λαμβάνουμε αναφορές. Τώρα, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Αυτή η Επιτροπή, σύν το χρόνο, όπως προκύπτει και από την παρακολούθηση του κοινοτικού δικαίου από την Κομισιόν, προκύπτει λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος τομέας προβλημάτων και ανησυχίας είναι το περιβαλλοντικό τομέας. Κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Αντιμετωπίζουμε συνεχώς το εξής πρόβλημα. Προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε το εξής σύστημα. Αν έχεις ένα παλιό δέντρο, μια παλιά καρυδιά, προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε. Αλλά μερικές φορές πρέπει να προλάβεις ότι κάποιος θα προσπαθήσει να καταστρέψει το δέντρο. Γιατί αν γίνει η καταστροφή είναι πολύ αργά. Και δυστυχώς πολύ συχνά είμαστε σε αυτή την κατάσταση σε σχέση με το περιβάλλον. Ερχόμαστε εκ των υστέρων. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε πιο υπέρ της πρόληψης. Ε, παρά να προσπαθούμε εκ των υστέρων να διορθώσουμε τα πράγματα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν ένα λεπτό και μετά ο κ. Χάμερστάιν Μίντς πάλι ένα λεπτό. Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρομαι ε, σε κάποια από τα στοιχεία που ανέφερε και η συγγήτρια Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής, ότι με μεγάλη μου χαρά να παρέμβω για να επιταχύνω την εργασία που γίνεται σχετικά με την καλύτερη πρόσβαση ε, των πολιτών ε, ε, σε ενημέρωση και σε διάφορα μέτρα που λαμβάνονται με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό αφορά όλα τα τμήματα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλα αυτά όπως και εκείνα τα οποία εφήγησαν στο σημείο 3 και 6 του σχεδίου της έκθεσης. Όσον αφορά τώρα τους ε, πίνακες συσχετισμού, αυτό το έχουμε θίξει στην ε, Κορεπέρ και στο Συμβούλιο σε ένα θέμα που χρήζει παρακολούθησης και θα ε, ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Το θέμα που αφορά μεμονωμένα άτομα, αυτό είναι δύσκολο να το λύσει Κομισιόν, γιατί το όλο θέμα ζημιώνει άτομα που σε πολλές περιπτώσεις ε, εξαρτώνται από νομικές ε, συνήθειες ε, στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το σημείο υπεριθμών 3, να σας πω ότι εξετάζουμε το κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρχει μια καλύτερη διαδικασία σχετικά με την ενημέρωση για διαδικασίες επί παραβάση και υπάρχει μια ε, τράπεζα ε, δεδομένων ε, που δεν διατίθεται στο Κοινοβούλιο σε οποιονδήποτε άλλο, είναι δικιά μα, αλλά δεν έχει και κανένα νόημα να διαδίδουμε πληροφορίε σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, τελειώσατε εσεί, τώρα ο κύριο Χάμερστάιν Μίντ. Ε, πρέπει να πω ότι αυτά που είπε ήταν πολύ σωστά σχετικά με την απλούστευση, την διαφάνεια. Όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, γιατί χωρίς αυτά οι επίπονες αυτές διαδικασίες ε, είναι πολύ κουραστικές. Ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο που έχει του θεματοφύλακα του αστιφύλακα αν θέλετε για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Κανοποιητικά όλα αυτά αλλά από την άλλη ε, πρέπει να υπάρχει και μια όθηση από τους πολίτες, από, τους κοινοβου... το κοινοβούλιο αν θέλουμε να προχωρήσουμε τα κοινωτικά προγράμματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Γόλης για την άψογη προετοιμασία της, ο συνήθως. Βλέπετε λοιπόν ότι χαίρεται ευρείας εκτίμησης και αναγνώρισης. Στις 12 Μαρτίου, 12 η ώρα, εκπνέει η προθεσμία για την ε, κατάθεση τροπολογιών. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, που καθυστερήσαμε τη συνεδρίαση. Όλες οι άλλες αναφορές από το, την ομάδα Β, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρθηκαν,